Buongiorno a tutti, se prendete posto, per favore lì, possiamo cominciare. Abbiamo una mattina molto intensa, diciamo, di contenuti. Λοιπόν, λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με την παρουσίαση από πλευράς της κυρίας Μπουρή του νέου κώδικα ο οποίος συνιστά το νέο ουσιαστικά νομοθετικό πλαίσιο στον τομέα των ηλεκτρονικών τηλεπικοινωνιών γενικά. Το θέμα αυτό εκκρεμεί εδώ και αρκετά καιρό, αρκετό καιρό. Το δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτός ο νέος ο κώδικας λοιπόν των τηλεπικοινωνιών στην ουσία συγκεντρώνει τις τέσσερις νομοθετικές προτάσεις που μας έχουν απασχολήσει τα τελευταία 5-6 χρόνια Όλοι γνωρίζουμε από αυτές τις νομοθετικές πράξεις από τότε που ελήφθησαν εν βασ περιπτώσει υπόψη μέχρι τώρα έχουν υπάρξει τεχνολογικές εξελίξεις βαρβές και εξελίξεις και σε επίπεδο κοινωνικό σχετικά με την χρήση και την εφαρμογή των τεχνολογιών για, στα πλαίσια της κοινωνίας. Είναι λοιπόν απαραίτητο να αντιμετωπίσουμε αυτό το νομοθετικό μέσο να δείξουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι διατεθειμένο να συνεργαστεί πλήρως. Έχουμε μία με μία μισή ώρα για την αντιμετώπιση, για τη συζήτηση αυτού του θέματος. Θα ήθελα να προτείνω την εξή μορφή. 10 με 15 λεπτά για την κυρία Μπιουρή και μετά ένας γύρος με παρεμβάσεις των συντονιστών ή των αναπληρωτών τους. Μια πρώτη απάντηση από πλευράς της κυρίας Μπυρή, έτσι ώστε να υπάρξει μια πρώτη αξιολόγηση και αμέσως μετά θα δώσω το λόγο στα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής μας. Λοιπόν, σας δίνω το λόγο πάνω σε ένα πραγματικά ιδιαίτερο θέμα. Καλημέρα λοιπόν σε όλους όσοι είστε εδώ σήμερα. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή που με καλέσατε εδώ σήμερα. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι εδώ από τότε που ανέλαβα τη θέση μου, που ήρθα στη θέση αυτή από το μήνα Ιανουάριο. Είναι μεγάλη τιμή επίσης για μένα να παρουσιάζω αυτήν την εν πολύ αναμενόμενη εδώ και καιρό πρόταση. Είναι τμήμα των προσπαθειών που κάνουμε εμείς στα πλαίσια της ε, εσωτερικής ψηφιακής αγοράς, της ενιαίας μάλλον ψηφιακής αγοράς. Έπρεπε να κωδικοποιήσουμε πολλές νομοθετικές πρωτοβουλίες και ρυθμίσεις, να τις απλουστεύσουμε και να κάνουμε και σημαντικές αλλαγές στα πλαίσια του ιδίου πλαισίου, έτσι ώστε τελικά να έχουμε έναν τηλεπικοινωνιακό κώδικα ο οποίος θα λειτουργήσει σαν πλαίσιο για την ολοκλήρωση της ψηφιακής αγοράς. Ελπίζω η συνεργασία που ξεκινάμε σήμερα να είναι μια καποφόρα συνεργασία. Το πλαίσιο αυτό σας ε, είναι και για σας καθοριστικό στα πλαίσια των εργασιών σας και ελπίζω να βρεθεί μια καλή λύση. Στα μέσα Σεπτεμβρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε το λεγόμενο Connectivity Package, το πακέτο συνδεσιμότητας. Θα σας παρουσιάσω τα μέτρα τα οποία περιλαμβάνει. Ε, πρώτον θα μιλήσουμε για τους λεγόμενους στόχους gigabit. Gigabit λοιπόν ε, δεν έχουμε την ψηφιακή αγορά που επιθυμούμε αν δεν έχουμε πραγματικά υπερσύγχρονη συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο σε όλη την Ευρώπη όχι μόνο στις πόλεις αλλά και στις περιοχές της υπαίθρου. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Δεν μπορούμε να χάσουμε λοιπόν αυτήν την δυνατότητα, από αυτήν εξαρτάται η ανταγωνιστικότητά μας και επίσης και η κοινωνική μας και η εδαφική μας συνοχή. Γι' αυτό ακριβώς λοιπόν παράγουμε ένα πλαίσιο το οποίο έχει σαν στόχο το 2025, έχει θα έλεγα ένα, ένα πολιτικό. Ε, θέλουμε όλοι να έχουν ε, ε, την επαρκή συνδεσιμότητα, ίσως να κατανεμηθεί δηλαδή σε όλη την Ευρώπη. Μιλάμε λοιπόν για τη συνδεσιμότητα για μια ανταγωνιστική ε, ψηφιακή ενιαία αγορά προς μια ευρωπαϊκή κοινωνία Gigabit. Οι ε, στόχοι αυτοί είναι συμπληρωματικοί με τους στόχους οι οποίοι έχουν ε, τεθεί και στα πλαίσια της ψηφιακής ατζέντα. Έχουν βέβαια και ένα πιο μακρό χρόνο για να αναπτυχθούν. Πώς θα μειώσουμε λοιπόν τις διαφορές που υπάρχουν, τι σημαίνει αυτό για τους πολίτες στην καθημερινότητά τους. Πρώτον, θα πρέπει να δούμε ότι οι βασικοί κοινωνικο-οικονομικοί, θα έλεγα, φορείς όπως σχολεία, τα hub των συγκοινωνιών, μιλάμε για μεγάλα κέντρα στα οποία συγκεντρώνεται μεγάλος αριθμός πολιτών και νέων παιδιών κτλ. Για αυτές τις περιοχές θέλουμε να έχουμε την καλύτερη δυνατή συνδεσιμότητα για να μπορούμε να συνεισφέρουμε και στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης με τον καλύτερο τρόπο. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά, να σας δώσω κάποια παραδείγματα. Αν έχουμε ας πούμε τέτοιου είδους gigabit συνδεσιμότητα, τότε μπορεί κάποιος να κάνει ε, ένα σκάνινγκ ε, μέσα μια σάρωση εικόνας ε, ή αντικειμένου σε 40 δευτερόλεπτα και όχι σε 20 λεπτά ή σε μισή ώρα. Επίσης και όταν ένας σερβερ σε μια επιχείρηση παρουσιάσει πρόβλημα μπορεί να διορθωθεί το ταχύτερο δυνατόν, χωρίς καθυστερήσεις. Δεύτερον, εμείς θέλουμε να έχουμε ε, κάλυψη 5G. Ε, ξέρουμε ότι υπάρχουν διαφορές ε, ανάμεσα στα επίπεδα κάλυψης σήμερα, ενώ το 5G είναι συνεχές ή ήρεμη διαδικασία. Έχουμε επίσης και τον ενδιάμεσο στόχο του 2020, η συνδεσιμότητα 5G να είναι διαθέσιμη σε εμπορικό επίπεδο τουλάχιστον σε μία μεγάλη πόλη κάθε φορά από το 2018 και μετά. αυτά όλα παράλληλα με αυτά που κάνουμε ε, για τις ε, ίνες μεταφοράς δεδομένων. Επίσης όλα τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά, όχι μόνο στις πόλεις αλλά και στην Ήπεθρο, να έχουν πρόσβαση σε συνδεσιμότητα τουλάχιστον 100 MB ανά δευτερόλεπτο. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι όλα τα νοικοκυριά θα έχουν ε, πρόσβαση στο ελάχιστο ε, ύψος συνδεσιμότητας ε, το οποίο θα είναι απαραίτητο για την οικογενειακή χρήση, τηλεοράσεις, τηλέφωνα και διάφορες άλλες εφαρμογές έτσι ώστε να μην υπάρχει ε, ένα κενό ψηφιακό ανάμεσα στις διάφορες περιφέρειες. Και οι τρεις αυτοί στόχοι σημαίνει ότι απαιτούνται δίκτυα υψηλής χωρητικότητας και γι' αυτό και το πακέτο αναδιάθρωσης των οδηγιών έχει ανάγκη και από επενδύσεις και θα επανέλθω σε αυτό αργότερα. Απαιτείται λοιπόν ε, μια νέα προσπάθεια συλλογική. Εμείς σαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή ελπίζουμε να συμφωνήσετε με τους στόχους αυτούς και σε πολιτικό επίπεδο και να καταστήσουμε αυτήν την κατάσταση πραγματικότητα. Υπάρχουν τρία μέτρα στο πακέτο αυτό. Το πρώτο το είπε και ο κύριος Γιούνκερ. Είναι το ελεύθερο Wi-Fi αυτό που ονομάζουμε σήμερα Wi-Fi for you, EU μάλλον. Αυτό θα πρέπει να καλύπτει βιβλιοθήκες, πάρκα, κεντρικές πλατείες, ε, κομβικά κτίρια στις πόλεις. Ε, ενθαρρύνουμε και στηρίζουμε τις τοπικές αρχές να το πραγματοποιήσουν όπου δεν γίνεται. Έτσι ώστε ο καθένας Wi-Fi ε, να δει πόσο επηρεάζει τη ζωή του. Η πρωτοβουλία αυτή και το είπε ο πρόεδρος Γιούνκερ δίνει την δυνατότητα να έχουμε και άλλη μία πραγματική απόδειξη του τι κάνει η Ευρώπη. Ελπίζω να προωθήσει την χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών, βλέποντας ποιες είναι οι ανάγκες με υψηλή ταχύτητα που διευκολύνει την καθημερινότητα το σύστημα αυτό θα, θα γίνει σιγά σιγά σε μικρούς χώρους από την αρχή. Τα χρήματα που θα απαιτηθούν δεν θα είναι πάρα πολλά, θα είναι απλό και μη γραφειοκρατικό. Ελπίζουμε το πρώτο Wi-Fi for You να είναι έτοιμο στο τέλος του 2017, έτσι ώστε να μπορέσει το σύστημα να λειτουργήσει ταχύτατα. Θα πρέπει ο κόσμος να μπορεί να το δει αυτό, να το επιλέγει όταν ανοίγει τα κινητά του τηλέφωνα στους δημόσιους χώρους που είναι διαθέσιμο. 130 εκατομμύρια για τρία χρόνια δεν είναι πάρα πολλά τα χρήματα, αλλά αν χρησιμοποιηθούν σωστά μπορούν συμβολικά να λειτουργήσουν θετικά. Θα μπορέσουμε λοιπόν να δώσουμε έτσι ε, συνδεσιμότητες σε 6 με 8 χιλιάδες τοπικές ε, κοινότητες. Αυτό σημαίνει ε, ότι πολλοί κόσμος θα ωφεληθεί από αυτό. Αυτό σημαίνει δηλαδή περίπου 40 με 50 συνδέσεις την ημέρα. Θα συνεχίσουμε την προσπάθεια αυτή για να πετύχει το μέσο αυτό γρήγορα δεν μπορούμε εμείς να αγνοήσουμε τις προσδοκίες των πολιτών και ε, θέλουμε και τη δική σας υποστήριξη για την πρωτοβουλία αυτή. Το δεύτερο τμήμα του πακέτου είναι το πρόγραμμα δράσης 5G. Εγώ αναφέρθηκα στην ανάγκη να υπάρχει ανεμπόδιστη πρόσβαση 5G σε ταχύτητες 5G. Έχουμε λοιπόν ένα πρόγραμμα δράσης το οποίο θα θέσουμε σε εφαρμογή ε, μέχρι το 2020 να πετύχουμε ε, το ε, στόχο αυτό και να δούμε τι συνέβη και με το 4G και να, πάρουμε τα, να βγάλουμε τα κατάλληλα συμπεράσματα. Εμείς έχουμε προτείνει ένα οδικό χάρτη για τη συνεργασία ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Νομίζω ότι αυτό το οποίο είναι το βασικό αυτό είναι ε, να ξεκαθαριστούν και να παραλληλιστούν όλοι οι οδικοί χάρτες και προτεραιότητες για να πετύχουμε ένα συντενισμένο τρόπο ανάπτυξης του 5G. Ε, θα συμπληρωθεί το φάσμα των συχνοτήτων από τις επιπλέον συχνότητες. Ε, ξέρετε ότι εργαζόμαστε για την πρόταση για τα λεγόμενα 700. Επίσης θέλουμε να ασχοληθούμε ε, και με κάποιες δοκιμές ε, συνεργασίας των σημείων αυτών στα οποία θα είναι διαθέσιμο το 5G έτσι ώστε να φτάσουμε στην ενιοποίησή του το ταχύτερο δυνατόν. Και τέλος, και αυτό είναι σημαντικό, ε, συνεργαζόμαστε με την βιομηχανία και τους ζητάμε να προωθήσουν το κοινό όραμα και τις κοινέ προτεραιότητες για ένα ενιαίο τρόπο 5G. Τέλος και είναι βασικό εδώ το θέμα για μας και για σας είναι ο κώδικας ε, των τηλεπικοινωνιών, ο Ευρωπαϊκός Ηλεκτρονικός Κώδικας και το Μπερέκ, ο κανονισμός Μπερέκ. Απαιτούνται 500 δις ε, την επόμενη δεκαετία ναι. Έχουν γίνει κάποιες εκτιμήσεις και από ό,τι φαίνεται ελείπουν στην παρούσα φάση 155 δις. Θα πρέπει να εξυγχρονιστούν οι κανόνες των τηλεπικοινωνιών έτσι ώστε αυτά τα 155 δις να έλθουν. Ο νέος αυτός κώδικας λοιπόν ενισχύει τις υπάρχουσες ρυθμίσεις για τον ανταγωνισμό αλλά υπογραμμίζουμε περαιτέρω τον ανταγωνισμό για επενδύσεις στα δίκτυα, έτσι ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι να έχουν ίδιες δυνατότητες. Ε, οι επιχειρήσεις αυτό το οποίο μας λέγουν είναι ότι απαιτείται νομική βεβαιότητα για να προχωρήσουν και προβλεψιμότητα. Γι' αυτό λοιπόν θα προωθήσουμε τις εμπορικές συμφωνίες, τις μορφές συγχρηματοδότησης ε, μειώνοντας την ανάγκη για ρυθμιστικές παρεμβάσεις. Θέλουμε εμείς να δημιουργήσουμε κάποιες προτεραιότητες έτσι ώστε να υπάρξουν επενδύσεις και από εναλλακτικού χρήστες θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για περαιτέρω διασυνδεσιμότητα διάφορα, ανάμεσα στα διαφορετικά κέντρα. Είναι το θέμα του φάσματος ε, των συχνοτήτων δύσκολο, αλλά είναι τμήμα του πακέτου το οποίο προτείνουμε. Νομίζω ότι τώρα έχουμε δημιουργήσει τη σωστή δυναμική και θα υπάρξει πρόοδος. Το Κοινοβούλιο υποστηρίζει ισχυρά τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέχρι τώρα και σας ευχαριστούμε γι' αυτό ε, και ε, νομίζω ότι θα πρέπει να συνεχίσετε να υποστηρίζετε και την πρόταση αυτή. Απαιτείται φυσικά και μεγαλύτερη προβλεψιμότητα για τις επενδύσεις, ελάχιστη περίοδος αδειοδότησης για την κατοχή τμήματος φάσματος θα είναι 25 ετία, και θα πρέπει επίσης το ταχύτερο δυνατόν να καθοριστούν οι ε, τομείς στις ναι. οποίες θα δραστηριοποιηθούν οι διάφορες επιχειρήσεις. Να υπάρξει ένα προβλέψιμο πλαίσιο, εν πάση περιπτώσει. Επίσης υπάρχουν ε, και τα θέματα της υποχρέωσης κάλυψης η αναπτύξη συστημάτων συνδεσιμότητας σε επίπεδο μικρής ε, διάστασης, σε μικρή διάσταση. Έχουμε νομίζω κάνει μια πρόταση αρκετά εξισορροπημένη, βασισμένη στις αξίες τις οποίες μέχρι τώρα έχουμε ακολουθήσει και ελπίζω να προχωρήσουμε γρήγορα. Τώρα τι σημαίνουν όλα αυτά για τους ε, καταναλωτές και τι προτείνουμε εμείς για τον ΠΕΡΕΚ, δηλαδή την ε, ρυθμιστική γενικά δυνατότητα που δημιουργείται. Ε, πρέπει οι χρήστες φυσικά να έχουν εμπιστοσύνη στα δίκτυα. Ε, είναι προϋπόθεση λοιπόν η προστασία των καταναλωτών εδώ και θα πρέπει να συνεχίσουμε να λαμβάνουμε μέτρα για την προστασία τους, όπου αυτό είναι απαραίτητο. Έχουμε αναβαθμίσει επίσης ε, και τις ε, ρυθμίσεις για την παροχή ε, καθολικού τύπου υπηρεσιών και για την δημιουργία θα αποσυρθούν ας πούμε οι τηλεφωνικοί θάλαμοι από τη μία, αλλά αυτό δεν θα είναι υποχρεωτικό για τα κράτη-μέλη, αλλά αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχει σύμβαση έτσι ώστε όλοι οι καταναλωτές να έχουν μια βασική δυνατότητα συνδεσιμότητας. Για να υποστηρίξουμε τους νέους κανόνες θα πρέπει να ανανεώσουμε αν θέλετε το υπάρχον θεσμικό σύστημα Και έχουμε το Μπερέκ εδώ, το οποίο συγκεντρώνει όλες τις ρυθμιστικές αρχές σε εθνικό επίπεδο ε, και νομίζω ότι μπορεί να λειτουργήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο στα πλαίσια της εξυπηρέτησης των κοινών μας στόχων και των δικαιωμάτων που έχουν ε, οι πολίτες ε, για την χρήση της συνδεσιμότητας. Λοιπόν, κλείνοντας, Πιστεύουμε ότι οι δυνατότητες στον τομέα της ψηφιακής αγοράς ε, δεν θα πρέπει να είναι για λίγους αλλά για όλους. Αυτός είναι ο βασικός μας στόχος. Γνωρίζουμε ότι το ευρύ φάσμα με υψηλές ταχύτητες έφτασε ήδη στο 70% των κατοικιών αλλά συγκεντρώνεται σε πυκνές αστικές περιοχές και μόνο το 28% των κατοικιών στην Ήπεθρο καλύπτονται. Αυτό δεν μπορούμε να το δεχτούμε, πρέπει να βρεθεί λύση. Οι προτάσεις αυτές νομίζω ότι θα τις επεξεργαστούμε καλύτερα μαζί σας και θα βρούμε λύσεις. Αν θέλουμε οι πολίτες ήδη από το 17 να ωφεληθούν, θα πρέπει να προχωρήσουμε και με την πρωτοβουλία Wi-Fi for You, και θα πρέπει να συζητήσουμε ακόμα περισσότερο μια εξυγχρονισμένη μορφή αυτού του κώδικα λοιπόν, ο οποίος τώρα βρίσκεται σε στάδιο μετάφρασης, έτσι ώστε γρήγορα να προχωρήσουμε. Ελπίζω να υπάρξει μια πολιτική συμφωνία στο τέλος του 2017. Αυτή είναι η φιλοδοξία την οποία έχουμε. Έχει σημασία <coughs> να κρατήσουμε την ταχύτητα που απαιτείται γιατί αλλιώς οι επιχειρήσεις μας δεν θα μπορέσουν να λειτουργούν με τις ταχύτητες που απαιτείται και δεν θα είναι τόσο ανταγωνιστικές. Εμείς θέλουμε το πολιτικό μας όραμα λοιπόν να γίνει πραγματικότητα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστούμε για αυτή την παρουσίαση που ήταν σαφέστατη και πληρέστατη. Σας διαβεβαιώνω ότι είμαστε πολύ έτοιμοι να ανταποκριθούμε σε αυτή την πρόκληση το Κοινοβούλιο και αυτή η Επιτροπή και όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα και τους φιλόδοξους στόχους που εμπεριέχονται στον κώδικα σήμερα στους συντονιστές Φερρυπίν ίσως ε, θα, καθοριστούν, ε, θα καθοριστεί ποιος θα είναι συγγητής για το πακέτο. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Και αν δεν γίνει σήμερα, στην επόμενη συνεδρία των συντονιστών, σίγουρα. Ξεκινάμε τις παρεμβάσεις των συντονιστών και μετά τις πρώτες απαντήσεις που θα δώσει η κυρία Μπιωρή και με άλλες παρεμβάσεις μετά. Συνάδελφε Κάριν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστούμε την Επιτροπή για αυτή την πρωτοβουλία. Όλοι την περιμέναμε. Επί μεγάλο χρονικό διάστημα, κανείς στην αίθουσα δεν αμφισβητεί ότι για να μείνει ανταγωνιστική η Ευρώπη και να ηγείται στον κόσμο, θα πρέπει να είμαστε δεμένοι με το διαδίκτυο, να υπάρχει συνδεσιμότητα. Τώρα θα αναφερθώ περισσότερο σε ανησυχίες παρά στα στοιχεία που ενθουσιάζουν και που είναι τα περισσότερα. Ποια είναι η ανησυχία μου. Να μην πέσουμε σε παγίδα. Να μην υποσχεθούμε κάτι που τελικά θα υλοποιηθεί. Wi-Fi for you ακούγεται καλό. Προσφέρουμε στον κόσμο δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο. 6.008 κέντρα σε 500 εκατομμύρια, ε, αγορά 500 εκατομμυρίων δεν τόσα πολλά και τα χρήματα που αναφέρατε για τη χρηματοδότηση δεν νομίζουμε ότι είναι αρκετά. Οι ιδέες καλές και άγιες, αλλά είναι εξίσου σημαντικό να είμαστε πραγματιστές στο τι υλοποιούμε και στο τι λέμε στον κόσμο, τι προσδοκίες δημιουργούμε. Αυτή είναι μια ανησυχία. Ο στόχος που δηλώσατε και το είπα τουλάχιστον πέντε φορές είναι να οριμάσει το περιβάλλον για επενδύσεις. Αυτό είναι πολύ κρίσιμο. Πρέπει να εξορροπήσουμε την ανάγκη των επενδυτών, δηλαδή να έχουν κέρδος, απόδοση της επένδυσης και από την άλλη την επιθυμία των καταναλωτών για πολύ καλές υπηρεσίες όσο πιο φθηνά γίνεται. Πολύ δύσκολο να επιτευχθεί, εύκολο να δηλωθεί, αλλά από τα λόγια στην πράξη είναι κάτι διαφορετικό. Εν γέννη η πρωτοβουλία είναι πολύ ευπρόσδεκτη. αν συμφωνούν και άλλοι συντονιστέ η ομάδα μου θα ενδιαφερόταν να επιλεγούν οι εισηγητές και να ξεκινήσουν ε, οι εργασίες το ταχύτερο δυνατόν. Ένα από τα βασικά στοιχεία του 5G είναι το φάσμα. Ξέρουμε ότι συζητείται η διανομή του φάσματος. Κανείς δεν πιστεύει ότι δεν χρειάζεται ανακατανομή του φάσματος για να υλοποιηθεί το 5G αλλά σε πολλά μέρη της Ευρώπης έχει ήδη διανεμηθεί το φάσμα και αυτό έχει δημιουργήσει πονοκεφάλους για τα κράτη-μέλη. Χρειάζεται εξισορρόπηση επιθυμιών με πρακτικές λεπτομέρειες. Δεν θέλω να πω κάτι αρνητικό. Εξαιρετική πρωτοβουλία. Από την ομάδα μας θα υπάρξει μεγάλη υποστήριξη. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές όμως να δούμε τι υποσχόμεθα και τι μπορούμε να υλοποιήσουμε το ταχύτερο δυνατόν. Αυτά και ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, συνάδελφε Κάριενς, συνάδελφε Ντανίκα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και εγώ πιστεύω ότι αυτό το πακέτο που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, την χάνει μεγάλη υποστηρίξεως στο Ευρωκοινοβούλιο. Θα ήθελα να πω ότι επιτέλους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας υπέβαλε ένα πακέτο για το 5G την τελευταία στιγμή για να μπορέσουμε να καλύψουμε την υστέρησή μας έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών και των χωρών της Ασίας, κυρίως έναντι της Νοτιού Κορέας. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να γίνει διαδικασία συντονισμού και να επιληθούν τυχόν διαφορές για την διανομή του φάσματος. ίσως το φάσμα, η κατανομή του φάσματος να είναι ένα θέμα. Ε, κυρίως ε, η διανομή του φάσματος για ε, πολιτικό, για χρήση από πολίτες και για χρήση από στρατιωτικές μονάδες. Λοιπόν, υπάρχει ένας ανταγωνισμός για την υλοποίηση του δικτύου 5G. Πρέπει να κινηθούμε γρήγορα. Μια άλλη πτυχή που θέλω να αναφέρω, το Wi-Fi for You, είναι ένα καλό πρόγραμμα, αλλά ο διάβολος κρίνεται ως συνήθως της λεπτομέρειας και ο μηχανισμός κατανομής, διανομής θα είναι πολύ σημαντικός, διότι η γενική διαδικασία μπορεί να υπονομευθεί πανεύκολα και δεν ξέρουμε αν αρκούν και τα χρήματα που διατίθεται. Το πρώτο βήμα είναι σημαντικό. Αν πετύχει το πρώτο βήμα, μπορούμε να περάσουμε σε μεταγενέστερο στάδιο. Πώς θα γίνει η διανομή λοιπόν είναι κάτι πολύ σημαντικό, διαφορετικά η διαδικασία δεν θα προχωρήσει καλά. Όσον αφορά τον κώδικα και τους κανόνες για τις τηλεπικοινωνίες, εγώ πιστεύω ότι υπερβολικές διατάξεις και ρυθμίσεις έχουν αρνητικό αντίκτυπο στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Αν αντικαταστήσει κανείς πρωινό δεν μπορεί ο κανονισμός να είναι φάρμακο γιατί είναι οι πολλοί κανονισμοί να διορθώσουν τα προβλήματα της εσωτερικής αγοράς. Δεν διάβασα πολύ προσεκτικά το έγγραφο, πρέπει να το παραδεχτώ. Αλλά βλέπω ότι αυξάνεται η εξουσία του Μπέρεκ και αυτό δημιουργεί κάποιες ανησυχίες για μένα. Διότι αυτό που πιστεύω είναι ότι πρέπει να είναι σαφής οι όροι, ποιος είναι υπεύθυνο γιατί ποιος θα έχει την ευθύνη για τους διάφορους διαγωνισμούς κλπ. Δεν θα πρέπει να υπάρχει αλληλεπικάλυψης στα καθήκοντα των διαφορών φορέων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να καταρτήσει μια στρατηγική και μια πολιτική. Και ο άλλος φορέας, ο Μπέρεκ, θα πρέπει να ασχοληθεί με τις πρακτικές πτυχές. όταν δεν κινείται σωστά η Μπέρεκ δημιουργούνται προβλήματα για τις χώρες. Το είδαμε αυτό στην, ε, στις τηλεπικοινωνίες τέταρτης γενιάς. Χρειάζεται Διπλασιάστηκε ο χρόνος που χρειαζόταν για την υλοποίηση του 4G. Το ήξερε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό τότε. Στο τέλος δεν πετύχαμε πολλά. Η Μπέρεκ δεν ήθελε να λάβει υπόψη το κόστος για την διανομή του φάσματος για ε, την, της τηλεπικοινωνίας τέταρτης δεν θέλουμε να επαναληφθούν αυτά. Πρέπει να είναι τα καθήκοντα σαφώς καθορισμένα. Και θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όσον αφορά το ποιο εκτελεί τι. Σας ευχόμεθα κατά τα άλλα κάθε επιτυχία και θα σας υποστηρίξουμε πλήρως. Εκτός μικροφώνου, Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω, όπως και άλλοι συνάδελφοι, ε, σας ευχαριστήσω για την παρουσίαση που κάνατε και που παρουσιάσατε το περιεχόμενο του πακέτου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα πρέπει να υπάρχει διασυνδεσιμότητα στην Ευρώπη πράγματι και έχουμε φτάσει στα όρια των ταχυτήτων ε, που μπορούμε να πετύχουμε. Οπότε ε, θα πρέπει να έχουμε καλύτερη κάλυψη της επικράτης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαι εισηγητής για, το, για τις τηλεπικοινωνίες και δεν μπορώ παρά να πω ότι ξεκινήσαμε με μεγάλες ιδέες κατά το παρελθόν και καταλήξαμε να υλοποιήσουμε το 10% των στόχων. Ήταν πολύ δύσκολο να ανταποκριθούμε στις δημιουργηθήσεις προσδοκίες. Πράγματι, γι' αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Να σταθμίσουμε τι μπορούμε να κάνουμε και τι υποσχόμεθα. Πράγματι, ο τομέας των τηλεπικοινωνιών χρειάζεται βεβαιότητα και ασφάλεια όσον αφορά την ομοθεσία και το ρυθμιστικό πλαίσιο. Ελπίζω ότι αυτό που θα παράξουμε θα είναι κατάλληλα προσαρμοσμένο και ευέλικτο, ώστε να μπορεί να προσαρμοστεί και ο τομέας με την τεχνική, τεχνολογική πρόοδο. Να μην χρειάζονται πολλές αλλαγές στο μέλλον δηλαδή. Επίσης είναι απαραίτητο να ενισχυθούν τα διάφορα δίκτυα διαβίβασης πληροφοριών και από την άλλη θα πρέπει να προσέξουμε ούτως ώστε τα χρήματα που θα χρησιμοποιήσουμε, τα δημόσια χρήματα, τα κρατικά χρήματα. Αυτά τα χρήματα λοιπόν να μην ε, καταλήξουν σε λάθος χέρια και να μην ε, πετύχουμε τους στόχους μας με αυτά τα χρήματα. Καμιά φορά είναι καλύτερο να μην τα κάνει όλα ο δημόσιος τομέας και να κάνει προσπάθειες ιδιωτικός τομέας. Άρα η χρηματοδότηση του κρατικού τομέα πρέπει να γίνει προσεκτικά. Πρέπει να είναι σαφής ο καθορισμός των ρόλων που παίζουν οι διάφοροι φορείς. Αλλιώς ίσως περιοριζόμαστε όσον αφορά την επίτευξη των στόχων με τους διαθέσιμους πόρους. Υπάρχουν πολλές διευθύνσεις και πολλοί φορείς πρέπει να εναρμονιστούν κατάλληλα και έτσι μπορεί να μπορούμε να κινηθούμε καλύτερα κυρίως για το πρόβλημα της διανομής του φάσματος. Σίγουρα πρόβλημα θα είναι η απόφαση για τη διανομή του φάσματος που θα γίνεται σε επίπεδο 100 μελών και μετά θίθεται πρόβλημα διασύνδεσης μεταξύ 100 μελών. Ευχαριστούμε για την εισαγωγή. πιστεύω ότι ο νέος κώδικας θα οδηγήσει σε ταχύτερη ανάπτυξη και ότι όλες οι δραστηριότητες που παρουσιάσατε εδώ σήμερα συμπεριλαμβανομένου και του Wi-Fi for You θα στηρίξουν τα δίκτυα εν γέννη και τις τηλεπικοινωνίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ εσάς. Συνάδελφε Κάλλας, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρότασή της. Από την πλευρά μας Καλωσορίζουμε αυτή την ενοποιημένη, την ενιαία προσέγγιση και έχουμε κάποιες ερωτήσεις για το φάσμα. Ξέρουμε ότι κατά το παρελθόν ήταν πολύ δύσκολο θέμα όσον αφορά τα 700 MHz και το φάσμα αυτό. Έχετε καλύτερα σχέδια τώρα για τη διανομή του φάσματος. Μετά για το Μπέρεκ. Πολύ καλό να υπάρχει ευρωπαϊκός έλεγχος και υποπτία διότι τώρα επικρατούν τα εθνικά συμφέροντα και κανείς δεν υπερασπίζεται τα ευρωπαϊκά κοινά συμφέροντα όσον αφορά την υλοποίηση των προτάσεων. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον ανταγωνισμό στην αγορά τηλεπικοινωνιών. Ευπρόσδεκτη η προσέγγιση. Έχω και μια ερώτηση. Βλέπουμε πολλές προσφορές πακέτων Οπότε οι εταιρείε τηλεπικοινωνιών δεν προσφέρουν απλώς τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, αλλά και άλλα προϊόντα. Το εξέταση αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη σύγκριση διαφόρων υπηρεσιών που παρέχονται και πώς καθορίζεται η αγορά και η εξουσία και η θέση της κάθε εταιρεία. Τώρα των υπηρεσιών σε σχέση με υπηρεσιών παρέχονται με διάφορου αριθμού τηλεφώνων, όπω και η υπηρεσία του 112. Στην πράξη, πώ λειτουργεί. Αν δεν υπάρχει δίκτυο, πάλι μπορεί κανεί να καλέσει τι υπηρεσίε ανάγκης έκτακτη ανάγκη. Αν δεν υπάρχει διαδίκτυο και η χερσαία διασύνδεση δεν παρέχει πρόσβαση στις υπηρεσίες ε, έκτακτης ανάγκης. Τι γίνεται. Δηλαδή δεν πρέπει να παρέχονται υπηρεσίε οι οποίε να μην είναι μόνιμε και σταθερέ και να συνηθίσει ο κόσμο κάποιε υπηρεσίε και μετά αν δεν υπάρχει διασυνδεσιμότητα να μην μπορεί να τι χρησιμοποιήσει. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίαση και προσβλέπουμε στη συνεργασία μαζί σα. Ευχαριστώ. Συνάδελφε Ρέμοντ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και από μένα ευχαριστήσεις προς την Επιτροπή για αυτή την παρουσίαση. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό εγχείρημα Ελπίζω ότι θα προχωρήσει καλά. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η τελευταία επισήμανση, θεωρώ, σε σχέση με τη διασύνδεση όσον αφορά το χώρο της υπαίθρου που δεν βαίνει καλώς. Πρέπει να πούμε ότι αποτύχαμε εδώ σε σχέση με την αγορά για την κάλυψη των αναγκών των χώρων της υπαίθρου με επιδόσεις όσον αφορά αυτό το δίκτυο. χρειάζονται ρυθμίσεις για να αποκατασταθούν τα πράγματα. Και είναι μεγάλο τμήμα της Ευρωπαϊκής Επικράτειας. Και έτσι πρέπει να δούμε αυτό το ψηφιακό κενό. Δεν μπορούμε να, το, να αφήσουμε αυτούς τους ανθρώπους να απομονωθούν. Γι' αυτό το χαιρετίζω όταν υπάρχουν κάποιες πρωτοβουλίες να ενισχυθεί η ρυθμιστική αρχή ε, πανευρωπαϊκά. Αυτή τη στιγμή με μια σωστή αποδοτική ρύθμιση μπορούμε να προχωρήσουμε. Εδώ βρίσκονται όμως πολλά συμφέροντα σε αντίθεση με αυτά τα οποία θα χρειαζόμασταν πανευρωπαϊκά αν ξεκινήσουμε από το δημόσιο συμφέρον. Και πρέπει να πούμε ότι σε σχέση με τις εθνικές ρυθμίσεις είναι κάποιες ρυθμίσεις ε, για το διαδίκτυο που δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί ότι επαρκούν από πλευράς εθνικού επίπεδου. Και είμαι υπέρ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαδραματίσουν ένα σημαντικό ρόλο. Τώρα, για το δίκτυο αυτό θεωρώ ότι είναι ένα πολύ σημαντικό εγχείρημα. Να κάνουμε λόγο για δημόσιο συμφέρον όταν πρόκειται για τα θέματα δημοκρατίας και πολιτικής. Μπορεί να είναι μικρότερο διαστάσεων το πρόγραμμα. Όμως θα πρέπει εδώ να δούμε και το θέμα της ασφαλτόστρωσης ε, οδών που δεν γίνεται ταυτόχρονα σε όλες τις διαδρομές. Εδώ κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε. Είναι λοιπόν επενέσιμη αυτή η προσπάθεια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Συνάδελφε Κάπελ, τελευταία παρέμβαση πλευρά ε, συντονιστών. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την εκπρόσωπη της Επιτροπής για τον προβληματισμό και τις προτάσεις. Αναμείναμε να ακούσουμε και φυσικά όλοι υποστηρίζουμε την διάσταση γίγα ε, και γνωρίζουμε τους στόχους που δεν είναι καινούργιοι ταχύτατο διαδίκτυο που πρέπει να επιτευχθεί. Όμως την υλοποίηση του ταχύτατου ταχαίως διαδικτύου τα κράτη-μέλη πρέπει και αυτά να δράσουν. Εδώ στην Αυστρία, στη χώρα μου, συζητάμε εδώ και χρόνια για το δισεκατομμύριο του ευρέως φάσματος ε, και πρέπει να εξευρεθούν κίνητρα και μηχανισμοί ώστε ενισχυμένα να δράσουν τα κράτη-μέλη και να κινηθούν προς μια ενιαία κατεύθυνση ώστε να επιτευχθεί το ταχύ ε, διαδίκτυο. Ταχύ διαδίκτυο και στον χώρο της υπαίθρου όταν κάνουμε λόγο για την κάλυψη της επικράτειας και για την διασύνδεσιμότητα και την ηλεκτρονική κινητικότητα ή mobility, χρειαζόμαστε και το χώρο της υπαίθρου αυτές τις διασύνδεσεις, όπως και στα κέντρα. Και αυτό θα σημαίνει και κάποιες ε, επιπτώσεις χρηματοοικονομικά. Και ιδιαίτερα με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων θα πρέπει να συντονιστούμε ώστε τέτοια προγράμματα να υποστηρίζονται προγράμματα δηλαδή για την επέκταση και ενίσχυση ταχαίως διαδικτύου, ταχύτητα του διαδικτύου και ευρω, φάσματο φάσματος και για τον χώρο της υπαίθρου και για τις τεχνολογίες που είναι διαθέσιμες. Ε, η Ευρώπη πολλά μπορεί να κάνει. Αν δεν θέλει να απολέσει τον ρόλο πρωτοπόρου στην τεχνολογία η Ευρώπη, θα πρέπει να δράσει. Πρέπει να σκεφτούμε για τις τεχνολογίες αυτές και να δράσουμε ταχύτατα. Και εδώ χρειάζεται καλή συνεργασία και συντονισμός με τις βιομηχανίες και τις επιχειρήσεις, να μην καθυστερήσουμε. Και όταν θέλουμε να προχωρήσουμε σε εναρμόνιση, πώς θα προχωρήσουμε όταν δεν θα υπάρχει ένα κοινό φάσμα συχνοτήτων και κοινών στόχων για παράδειγμα στο τρένο όταν κινείται κανείς και περνάει ακόμα και από την Φραγκφούρτη ή άλλες πόλεις πολλές φορές δεν υπάρχει η διασφάλιση αυτής της ε, διασύνδεσης και εδώ πραγματικά συμφωνώ με τις ε, προτάσεις ε, και χρειάζεται εδώ τα ε, εκατομμύρια που αναφέρθηκαν δεν είναι ε, πολλά και όσον αφορά τις τοπικές κοινότητες για να διασυνδεθούν μέχρι το 2020 δεν φτάνουν αυτά τα χρήματα, 120 εκατομμύρια. Έχουν προαναγγελθεί σε σχέση με την, ε, τον ανταγωνισμό και της, ε, την ενίσχυση εδώ ένας ανταγωνισμός λέει των πόλεων. Εδώ θα πρέπει να μεριμνήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην υπάρξει ένας αθέμητος ανταγωνισμός και το υποστηρίζω να μπορέσουν οι κοινότητες ε, σε σχέση με τέτοιες δυνατότητες ε, να βρίσκονται σε ισότιμο πεδίο, σε ίση βάση. Αυτό ίσως μπορείτε να το εξετάσετε. Αν είναι δυνατόν να προχωρήσουμε μια χιονοστιβάδα επενδύσεων θα απαιτηθεί όχι μόνο για την βιομηχανία αλλά και για την αυξημένη ασφάλεια και όσον αφορά και την ασφάλεια των ρυθμίσεων και της ρυθμιστικής αρχής. Εδώ θα πρέπει να ε, γίνουν τα πράγματα σε ένα αυστηρότερο πλαίσιο για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ακούσαμε τον πρώτο γύρο παρεμβάσεων τα προβλήματα, ανησυχίες. Να σας δώσω αμέσως το λόγο, κυρία Μπέρι, να δώσετε απαντήσεις, ένα πρώτο γύρο απαντήσεων. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους τους συντονιστές για την υποστήριξή τους. Αυτό που ακούσαμε δείχνει ότι έχουμε τα καλά στοιχεία, τα σωστά στοιχεία στο πακέτο. Ακούσαμε κάποια ερωτηματικά, κάποιες ανησυχίες για το αν έχουμε εξισορροπήσει τα πάντα σωστά. Όσον αφορά το Wi-Fi for EU, κύριε Κάρενς, πρέπει να είμαστε πραγματιστές, διότι δεν έχουμε και πάρα πολλά χρήματα και σωστά, την Νίτσα, είπατε ότι ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες σε κάποιο βαθμό. Πρόθεση είναι να αυξήσουμε δυνατότητε, όχι να επιφέρουμε επανάσταση. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό με 120 εκατομμύρια. Ποια είναι η ιδέα, ο κόσμος να δει στην πράξη πώς λειτουργούν όλα αυτά και ελπίζουμε ότι αυτό θα σημάνει ότι θα δημιουργηθεί ζήτηση και όπως είπα μπορούμε να αρχίσουμε τη διαδικασία. Λοιπόν, 120 εκατομμύρια σε τρία χρόνια δεν είναι αρκετά, αλλά το πρακτικό κόστος των μονάδων που χρειάζεται για το Wi-Fi δεν τόσο πολλά. 20.000 ε, αναμονά θα δίνουμε. Περίπου 200 ευρώ κοστίζει για εσωτερική μονάδα και 500 για εξωτερική μονάδα και από αυτές τις μονάδες μπορεί να εξυπηρετείς πολλούς. 50 χρήστες ε, κάθε φορά που χρησιμοποιούν την μονάδα. Δεν είναι τεράστιο ποσό, αλλά αν το χρησιμοποιήσουμε συνετά μπορούμε να έχουμε σοβαρά αποτελέσματα. Όπως είπατε κύριε Νίτσε, μπορεί να αποτελέσει απαρχή αν ξεκινήσουμε την προσπάθεια, ίσω να αντλήσουμε και άλλα χρήματα στο μέλλον. Πρέπει να δείξουμε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σωστά και καλά τα 120 εκατομμύρια. Πώ, νομίζω, δύο πράγματα μπορούμε να κάνουμε. Πρώτα απ' όλα, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο πώ συνεργαζόμαστε με τα κράτη-μέλη και τι τοπικέ αρχέ. Χρειάζεται δίκαιη κατανομή, που ανέφεραν αρκετά μέλη, αλλά πρέπει να εξασφαλίσουμε και την ποιότητα ε, των υπηρεσιών που παρέχονται. Να είναι υψηλή ποιότητα δηλαδή θα πρέπει όσοι εφαρμόζουν τα ε, μέτρα ασχοληθούν και με τις λειτουργικέ δαπάνες και τελικά να είναι ποιοτικές υπηρεσίες που παρέχονται. Όσον αφορά την αποτελεσματικότητα, επανέρχομαι σε αυτά που προανέφερα. Πρέπει να είμαστε απλοί και γρήγοροι. Αν μπορούμε με ένα σύστημα δελτίων ούτως υπήν, δεν θα είναι τόσο μεγάλη αξία τους, 20.000 ανακοινότητα, αλλά θέλουμε γρήγορο και αποτελεσματικό σύστημα. Και γι' αυτό βασιζόμαστε σε εσά όταν θα συζητήσουμε την πρόταση. Να γίνει αυτό που ώστε να οδηγεί ε, σε ε, πρόσθετη, προστιθέμενη αξία, να δώσουμε μειώθηση στο όλο πρόγραμμα και τελικά να δώσουμε ποιοτικά προϊόντα στους χρήστες. Για τις επενδύσεις βέβαια, σωστά είπατε, ότι από τη μια πλευρά χρειαζόμαστε παραπάνω επενδύσεις, αλλά χρειαζόμαστε και καλή σχέση κόστου αποδοτικότητας για, τους, για τις υπηρεσίες που παρέχονται στους πολίτες, το έχουμε υπόψη. Υπάρχουν κάποια σημάδια σύμφωνα με τα οποία οι καταναλωτέ είναι πρόθυμοι να πληρώσουν για την ποιότητα, αλλά λογικέ τιμέ για την ποιότητα. Δεν θέλουν να πληρώσουν υπερβολικά τιμήματα για την ποιότητα, αλλά αυτό είναι μία από τι λεπτομέρειε που πρέπει να εξετάσουμε. Δηλαδή, πώ θα πετύχουμε τη σωστή ισορροπία, ούτω ώστε τηλεπικοινωνίε και οι φορείς που τι παρέχουν έχουν αρκετά χρήματα για επενδύσει, αλλά να παρέχουν την ποιότητα σε λογικέ τιμέ στους καταναλωτέ για το φάσμα. Σωστά το είπατε. Έχουμε θέματα ε, κληρονομιάς του υπήν όσον αφορά το φάσμα. Δεν θα πρέπει όμως να κολλήσουμε εκεί. Ε, όπου έχουν γίνει σφάλματα πρέπει να τα διορθώσουμε. Όσον αφορά το ερώτημα τη κύρια Κάλλα, δεν έχω μαγικό ραβδί, ούτω ώστε να τα διορθώσω όλα και να πω ότι αυτή τη φορά θα είναι εύκολα τα πράγματα. Δεν μπορώ να το πω αυτό, θα είναι δύσκολα. Όταν ήρθε εδώ ο Επίτροπο Έτιγκερ, είπε ότι πρέπει να συνεργαστούμε στενά με τη βιομηχανία, ούτω ώστε και αυτοί να διαβιβάσουν το μήνυμα στα κράτη-μέλη. Δηλαδή ότι χρειαζόμαστε, πρέπει να γίνουν όλα αυτά καλύτερα. Αυτό ήταν λογικό. Θα πρέπει και τα κράτη-μέλη να κάνουν αυτό που πρέπει, να παίξουν το ρόλο του στο παιχνίδι. Αλλά στο τέλο οι προτάσει μα είναι καλά εστιασμένε επί συγκεκριμένων θεμάτων για ε, το τι θέλουμε να πετύχουμε. Αν κάνουμε τη διαφορά, εκεί μπορούμε να δημιουργήσουμε τα προβλήματα, ε, συγγνώμη, να λύσουμε τα προβλήματα που έχουμε κληρονομήσει και από το παρελθόν. Το Μπέρεκ, ε, ε, αναφερθήκατε στο στον προβληματισμό τη εξουσία που έχει. Στην Μπέρεκ έχουμε μία ομάδα με τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες και θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις γνώσεις. Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο καθορίζουν το νομοθετικό πλαίσιο καθορίζονται γενικοί στόχοι, πώς θέλουμε να λειτουργήσει το σύστημα, θα υπομειστεί τις τη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά υπάρχει μια ανάγκη οι ρυθμιστικοί να εργαστούν μεταξύ τους, να ανταλλάξουν εμπειρίε. Και επί τη βάση αυτών ελπίζουμε ότι θα αποφύγουμε τις καταστάσεις που περιγράψατε στο μέλλον. Αλλά δίκαιο έχετε, απόλυτο δίκαιο. Πρέπει επακριβώ να τα καθορίσουμε αυτά. Το προβλέπει και η νομοθεσία. Να καθορίσουμε επακριβώ ποια θα είναι τα καθήκοντα των διαφόρων φορέων και θα πρέπει και να υπάρχουν και τα ελεγκτικά πλαίσια τα κατάλληλα. Κυρία Κάλλας, άλλο ερώτημα για την ομαδοποίηση των προϊόντων, πακέτων προϊόντων που αγοράζουν καταναλωτέ. Σωστά είπατε, ίσω να υπάρχουν θέματα ανταγωνισμού που προκύπτουν από αυτό. Ο τρόπο που το είδαμε εμεί το θέμα αυτό των πακέτων ήταν να το λάβουμε υπόψη στους κανόνες περί καταναλωτών. Δηλαδή επεκτείνουμε τους κανόνες περί καταναλωτών για να ισχύουν και για πακέτα υπηρεσιών και προϊόντων. Και αυτό θα επηρεάσει θετικά την κατάσταση. Το εξετάσαμε και καταλήξαμε συγκεκριμένη απάντηση όσον αφορά τους κανόνες περί τελικού χρήστου για την πρόσβαση στα, στους αριθμούς ε, έκτακτης ανάγκης και πώς θα λειτουργήσει στην πράξη ανάμεσα σε αυτούς που χρησιμοποιούν το σύστημα με αυτού του είδου του ειδικού αριθμού και αυτού που δεν το χρησιμοποιούν. Προσπαθήσαμε να πετύχουμε μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου στο θέμα, αν δείτε τι λεπτομέρειε τη προτάσεις. Θέλαμε να εξασφαλίσουμε ότι όλοι εκείνοι που χρησιμοποιούν του αριθμού, όχι μόνο οι παραδοσιακοί φορεί, αλλά και άλλοι οι νέοι φορεί, ότι θα πρέπει να παρέχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες ανάγκες και έχουμε και μηχανισμό διαφύλαξης ούτως ώστε να αντιμετωπίσουμε προβλήματα διαλειτουργικότητας να προκύψουν. Για εκείνους που είναι ανεξάρτητοι από αριθμό, που δεν χρησιμοποιούν τους αριθμούς ειδικού, έχουμε μηχανισμό διαφύλαξης, εάν χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί. Καλύπτεται. Η Επιτροπή θα συζητήσει λεπτομερέστερα το θέμα. Αν αυτός ο τρόπος που προτείνουμε είναι επαρκής ή όχι. Αυτό προτείναμε εμείς. Κύριε Ρεϊμούν, Αναφερθήκατε στη σημασία της διασυνδεσιμότητας στην Ήπεθρο, υποστηρίξτε το Wi-Fi, μην ξεχάσετε ότι έχουμε και το βασικό πακέτο διασυνδεσιμότητας στις ε, καθολικές υπηρεσίες. Εξετάστε τις λεπτομέρειες, δηλαδή τι έχουμε στο πακέτο αυτό. Ελπίζουμε ότι πετύχαμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ των βασικών υπηρεσιών. Είναι πολύ σημαντικά αυτά και για την Επιτροπή σας, δηλαδή οι βασικές υπηρεσίες να είναι προσβάσιμες στη σπάση. Κυρία Κάπελ, απάντησα κάποιες από τις ερωτήσεις σας. Αναφερθήκατε στο κόστος του Wi-Fi for you και τι όφελος θα δώσει. Υπογραμμίσατε ότι θα πρέπει και τα κράτη-μέλη να συνδράμουν και ευχαριστούμε και για την υποστήριξη που μας δώσατε για τις τηλεπικοινωνίες πέμπτης γενιάς. Ελπίζω κυρία Πρόεδρε να κάλυψα κάποιες από τις ερωτήσεις. Ναι, μάλιστα. Ευχαριστώ. Πιλάρ Δεκαστήγιο. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτή την παρουσίαση στη δική μας Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Πολύ λίγα έχω να προσθέσω, διότι είναι μια πρώτη συζήτηση με παρουσίαση αυτή. Οι συντονιστές είδαν γενικά με μια ανασκόπηση με απόψεις που συμπίπτουν σε μεγάλο βαθμό και μικρές διαφοροποιήσεις επί των μεγάλων θεμάτων και τώρα αυτό που πρέπει να γίνει είναι το νωρίτερο δυνατό να μπορέσει το Κοινοβούλιο να ξεκινήσει τις ε, κοινοβουλευτικές ε, διαδικασίες. Έχουμε προκλήσεις μεγάλης εμβέλειας μπροστά μας. Δεν μπορούμε να καθυστερήσουμε και να επεκτείνουμε την λήψη απόφασης ώστε αντικειμενικά να δημιουργήσουμε το ψηφιακό εκείνο πλαίσιο και περιβάλλον για να προχωρήσει η ενιαία ψηφιακή αγορά που έχει κέρια σημασία ώστε η οικονομία να μπορέσει σε παγκόσμιο πλαίσιο να είναι αποτελεσματική. Σε αυτό το πλαίσιο η διασυνδεμότητα είναι ο άξονας, η σπονδυλική στήλη όπως εξηγήσατε εσείς και λίγα μπορούν να προσθεθούν. Ουσιαστικά δεν θέλω να αναλώσουμε περισσότερο χρόνο. Το Κοινοβούλιο πρέπει να ξεκινήσει το δυνατόν νωρίτερα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον πλαίσιο να μπορέσει να κάνει και το Κοινοβούλιο σημαντικές συνεισφορές και παρεμβάσεις στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και χαίρομαι που άκουσα από τους συντονιστές των κοινοβουλευτικών ομάδων ότι γενικά ως γραμμή κίνησης έχουμε μια θετική αξιολόγηση αυτής της πρότασης της Επιτροπής που χωρίς αμφιβολία θα διευκολύνει τη συζήτηση και τις διαβουλεύσεις στο Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ και συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Κύριε Νάτρυπ, ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ καλή η πρόταση αυτή το ίντερνετ για όλους, γιατί πραγματικά πρέπει να αντιμετωπιστεί το θέμα των διαφορών κάλυψης στα πλαίσια της προϊούσας ψηφιοποίησης. Αυτό θα δημιουργήσει και καλύτερη ενιαία αγορά, θα προστατεύσει την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, θα προστατεύσει τους καταναλωτές. Νομίζω λοιπόν είναι πάρα πολύ καλή ιδέα αυτή το να προσπαθήσουμε και στη δική σας πρωτοβουλία Wi-Fi for EU να υπάρξει αποτέλεσμα. Αυτό είναι κάτι που θα δημιουργήσει και επιχειρήσεις και δυνατότητες για τους καταναλωτές. Η αλήθεια είναι βέβαια σε διασυνοριακές περιοχές ε, οι κλήσεις από τη μία χώρα στην άλλη ακόμα και αν είναι ανάμεσα σε γείτονες θα συνεχίσουν να κοστίζουν. Είναι καλό που αυξάνεται εν και αναπτύσσεται η ψηφιακή βιομηχανία ε, και η εσωτερική αυτή διασυνδεσιμότητα είναι καθοριστική και για άλλες επιχειρήσεις εκτός ψηφιακού τομέα για καινούργιες επιχειρήσεις που θα χρησιμοποιήσουν τις δυνατότητες που δίνει η ψηφιοποίηση και ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε λοιπόν ότι θα πρέπει να μεγιστοποιήσουμε τις επενδύσεις που θα γίνουν στον τομέα αυτό και να δώσουμε χώρο στις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν και να είναι ανταγωνιστικές. Οι ρυθμιστικές παρεμβάσεις δεν βοηθούν πάντα και γι' αυτό θα πρέπει να δούμε ότι ε, δεν θα πρέπει να υπάρξουν περαιτέρω ρυθμιστικές παρεμβάσεις πρέπει να προσπαθήσουμε να διαμορφώσουμε ένα ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού. Το θέμα της προβλεψιμότητας για τις επενδύσεις και τις βιομηχανίες είναι σημαντικό και είναι σωστό αυτό που είπατε ότι έχουμε κάνει κάποια λάθη και άλλες ήπειροι έχουν προχωρήσει πιο γρήγορα και η καινοτομία δημιουργείται σε άλλες ήπειρους γιατί εμείς να δεχόμαστε παθητικά την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί ότι οι μηχανές χτίζονται στην Άπο Ανατολή, το περιεχόμενο και το λογισμικό στη ΣΥΠΑ και εμείς κάπου πουθενά. Η κυρία Γκρίφιν. Ευχαριστώ Πατρίσια, ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η παρουσίασή σας ήταν πραγματικά αισιόδοξη και πράγματι θα υποστηριχθείτε πλήρως. Εγώ εκπροσωπώ την βορειοδυτική Αγγλία που περιλαμβάνει τις πόλεις του Μάντσεστερ και του Λίβερπολ και τις περιοχές της Κάμπρια και του Λάνκασαερ. Και πολλές από τις κοινότητες αυτές έχουν ε, μεν πρόσβαση σε υψηλής ταχύτητας διαδίκτυο αλλά οικονομικά αυτό έχει δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα. Αναφερθήκατε επίσης και στα θέματα προστασίας της υγείας και στην πρόνοια την ιατρική. Νομίζω ότι μπορούμε χρησιμοποιώντας την ψηφιοποίηση να διευκολύνουμε την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και να βοηθήσουμε να μην απομονώνονται κάποιες περιοχές. Αυτό νομίζω ότι και μέσω της παροχής καθολικού τύπου υπηρεσιών ε, θα πρέπει να ε, προχωρήσουμε και στον τομέα της ε, νομικής ασφάλειας και βεβαιότητας. μία μικρή παρατήρηση. Όλοι θα πρέπει να έχουν επαρκή διασυνδεσιμότητα και θα πρέπει όμως να βοηθήσουμε και τους καλύτερους στον τομέα. Προφανώς θα πρέπει να έχουμε πολιτική πρόθεση όλοι οι πολίτες να είναι οι πρώτοι, να είναι οι καλύτεροι. Επίσης είπατε στις απαντήσεις που δώσατε στις ερωτήσεις ότι οι τοπικές κυβερνήσεις παίζουν σημαντικό ρόλο, οι τοπικές αρχές. Ε, πράγματι μπορεί να ωφεληθούν και από τα διαφορετικά ταμεία γι' αυτό, αλλά νομίζω ότι και σε επίπεδο ε, σκέψης θα πρέπει να δούμε τι μπορεί να κάνει τώρα η τοπική αυτοδιοίκηση. Το Ηνωμένο Βασίλειο ελπίζω να συνεχίσει ε, να συμμετέχει στη διαδικασία αυτή και το hashtag wifi for είναι κάτι το οποίο αυξάνεται συνεχώς. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την Επιτροπή για την παρουσίασή της. Νομίζω ότι είναι σωστό να πει κανείς ότι η υποδοχή της πρότασης είναι μια θετική υποδοχή. Και αυτό για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί πράγματι υπάρχει ένα σημαντικό βήμα το οποίο πρέπει να γίνει. Και δεύτερον, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, κατά κάποιο τρόπο ε, υπόσχεται σε όλους τα πάντα Γι' αυτό λοιπόν όλοι γνωρίζουμε ότι στην πραγματικότητα θα πρέπει να βάλουμε προτεραιότητες. Και γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε ηγέτες σε πλαίσιο χρήσης του 5G, του 5G. Αυτό θα βοηθήσει την ευρωπαϊκή οικονομία να παραμείνει ανταγωνιστική θα πρέπει να δούμε λοιπόν ότι ναι μεν πρέπει να προστατεύσουμε τα συμφέροντα των χρηστών, των καταναλωτών, αλλά και πώς εμείς με τις ρυθμίσεις μας θα προσελκύσουμε καινοτόμες επενδύσεις. Ε, είναι καλό επίσης να μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είτε σήμερα είτε αργότερα για το τι ε, πρέπει να κάνουμε από εδώ και πέρα σε επίπεδο προτεραιότητας. Γιατί αν προσπαθήσουμε να τα κάνουμε όλα τότε σημαίνει ότι δεν έχουμε προτεραιότητες και πολλές φορές ε, έχουμε και συγκρούσεις συμφερόντων. Σαν παράδειγμα έχει σημασία το ταχύτερο δυνατόν να δημιουργήσουμε ακριβώς τον ελεύθερο χώρο στο φάσμα συχνοτήτων για την κινητή τηλεφωνία και τα δεδομένα. Έχει μεγάλη σημασία να το κάνουμε αυτό και έχει μεγάλη σημασία επίσης να μπορέσουμε να μοιραστούμε δίκτυα και ε, σε επίπεδο οπτικών ινών. Όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν, αλλά σε επίπεδο προτεραιότητας. Κάποια είναι πιο επίγοντα από άλλα Δεν ξέρω αν ξεκινάμε με τη λογική ότι όλα αυτά θα πρέπει να είναι δωρεάν, γιατί ε, αυτό μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. Ευχαριστώ κύριε Χόκμαρκ. Ο κύριος Ρόντε. Ελπίζω να μπορέσω να πω και εγώ τη γνώμη μου γύρω από το θέμα αυτό, συγχαίροντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το σχέδιο το οποίο έχει Νομίζω ότι θα πρέπει με τα μέσα τα οποία προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιδιώξουμε τους στόχους τους οποίους αναφέρθηκε. Υπάρχουν δύο πράγματα στα οποία θα ήθελα να σταθώ. Καταρχάς, αν θέλουμε να έχουμε ένα λειτουργικό 5G ε, ε, το ταχύτερο δυνατόν, σε ένα λογικό βέβαια χρονικό διάστημα, ε, ποιο θα είναι το χρονοδιάγραμμα θα πρέπει να είμαστε φυσικά, για να το πετύχουμε αυτό, πολύ πιο φιλόδοξοι σε σχέση με την χρήση και τις ρυθμίσεις στο φάσμα των συχνοτήτων. Και να δούμε ακριβώς τι θα γίνει επίσης και με την χρήση των ε, συχνοτήτων άνω των 700 MHz και με τη χρήση των συχνοτήτων κάτω από το, από το συγκεκριμένο αυτό στόχο. Ένα άλλο βασικό πρόβλημα εδώ είναι ότι μας λείπουν χρήματα για τη δημιουργία των υποδομών. Απαιτείται να επενδύσουμε σε επίπεδο υποδομών πολύ περισσότερο από ό,τι το κάνουμε τώρα. Γι' αυτό λοιπόν το Wi-Fi for you είναι κάτι το οποίο μπορεί να λειτουργήσει σαν παράδειγμα και νομίζω ότι το να αφήσουμε βέβαια όλα αυτά να αναπτυχθούν σε επίπεδο α, επικουρικότητας δεν αρκεί. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε περισσότερες πιστώσεις έτσι ώστε να μπορέσουμε να μετατρέψουμε και τα διαρθρωτικά μας ταμεία γιατί ξέρετε ότι έχουμε ένα υψηλό επίπεδο πιστώσεων και θα πρέπει τα διαρθρωτικά αυτά ταμεία να λειτουργήσουν σε επίπεδο ε, υποδομών για την Ευρώπη και στην ενέργεια και στους σιδηροδρόμους και στα διαδίκτυο έτσι μόνο θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην Ευρώπη. Πρέπει λοιπόν να είμαστε πιο φιλόδοξοι από ό,τι σήμερα σε σχέση με την συνδεσιμότητα. Πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορέσει να λειτουργήσει ε, σαν αναπτυξιακό κέντρο για την Ευρώπη και έτσι να δημιουργήσει και θέσεις απασχόλησης θα πρέπει εμείς να προσπαθήσουμε να δούμε τις κατηγορίες με διαφορετικό τρόπο από ό,τι σήμερα. Αλλά για να γίνουν όλα αυτά απαιτούνται χρήματα. Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να εναρμονίσουμε ε, τις ε, δυνατότητες τις οποίες έχουμε και ιδιαίτερα να χρησιμοποιήσουμε με σωστό τρόπο ε, τις δυνατότητες που μας παρέχουν οι συχνότητες. Σας ευχαριστώ κύριε Ρώτε και στο φόρου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πραγματικά θα ήθελα να αρχίσω ευχαριστώντας την αναπληρωτή Γενική Διευθύντρια της Γενικής Διεύθυνσης για την εξαιρετική παρουσίαση, αλλά πολύ περισσότερο γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ίσως από τις λίγες φορές δείχνει να βρίσκεται ένα βήμα πιο μπροστά να υλοποιεί θέσεις και απόψεις του Ευρωκοινοβουλίου και να δημιουργεί αυτή ένα πολύ ωραίο όραμα για την ψηφιακή οικονομία που απαιτεί όμως υλοποίηση. Πολλές φορές τονίσαμε ότι πλέον το διαδίκτυο είναι βασικό ανθρώπινο δικαίωμα. Και αυτό το βασικό ανθρώπινο δικαίωμα δεν μπορεί να το στερείται κανένας. Και υπάρχει μεγάλο χάσμα και δυσμενής διάκριση και μεταχείριση όταν υπάρχουν περιοχές μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε αγροτικές είτε απομονωμένα νησιά, τα οποία οι νέοι άνθρωποι ιδιαίτερα δεν έχουν το δικαίωμα και τη δυνατότητα να κάνουν τη χρήση του διαδικτύου. Είτε από οικονομική αδυναμία, είτε γιατί ποτέ το διαδίκτυο δεν μπορεί να φτάσει σε αυτέ τι περιοχέ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ορθά μπορεί να διαθέτει πολλά δισεκατομμύρια και σε άλλε περιοχέ του κόσμου για να μπορέσει να τι αναπτύξει και να τι αναβαθμίσει ποιοτικά. Είναι αδιανόητο τι δικέ τη περιοχέ μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο μέχρι σήμερα να τις κρατεί έξω από την πρόσβαση σε αυτό το βασικό δικαίωμα που είναι το Wi-Fi. Άρα υιοθετώ πλήρω την θέση και την άποψη για το Wi-Fi for you. Όμω χρειάζονται χρήματα. Διαθέτουμε πολλά δισεκατομμύρια σε αμφιβόλο αξία έργα και απόδοση πολλέ φορέ και το να δίνουμε μόνο 120 εκατομμύρια για τρία χρόνια για το Wi-Fi for you πιστεύω ότι είναι ε, αδιανόητο και θεωρώ ότι έγινε το πρώτο βήμα και πρέπει αυτά τα κονδύλια να τα επαξίσουμε. Γιατί αν έχει ένα τομέα που η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να κάνει τη διαφορά, μια Ευρωπαϊκή Ένωση που ουσιαστικά περικλείεται από χίλια δυο προβλήματα και τη ασκείται διαρκώ κριτική, είναι η ψηφιακή οικονομία. Και αν υλοποιήσει αυτό το όραμα για Wi-Fi for you στην πράξη και όχι μόνο θεωρητικά, θα κάνει τη διαφορά. Για μένα είναι αδιανόητο ένα ιδιώτη, ο ιδρυτή του Facebook, ο Μάρκ Ζούγκεμπεργκ, να διακηρύττει ότι μπορεί να καλύψει περιοχές που δεν έχουν Wi-Fi με δωρεάν Wi-Fi και να δυνατεί να το πράξει η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα θεωρώ ότι το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρώπης είναι η ίδια ψηφιακή οικονομία και το κέρδος θα είναι πολλαπλάσιο. Εγώ έχω να κάνω και μια ανησύγηση. Όπως πολύ ορθά το Ευρωκοινοβούλιο ψήφισε μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δοθεί κάρτα στου νέου με το e-trail για να μπορούν να έρθουν σε επαφή με, την, με ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύω ότι αυτή η κάρτα για δωρεάν Wi-Fi, αν μπορούσε να δοθεί στου νέου, για να μπορέσουν να έχουν πρόσβαση στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί είναι πιο εύκολο να έχει πρόσβαση με το ίντερνετ για να δει τι λειτουργίε και το έργο που παράγει η Ευρωπαϊκή Ένωση, από το να πάρει το τρένο και να μπορέσει να γνωρίσει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα θα μπορούσαμε να υλοποιήσουμε κάτι ανάλογο για του νέου ανθρώπου. Εμεί στηρίζουμε από την αρχή μέχρι το τέλο για να μην τα αναλύσω όσα αναφέρθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα τα στηρίξουμε όμως η απέτηση είναι ότι τα 120 εκατομμύρια είναι πολύ λίγα, πρέπει να επαυξηθούν άμεσα και οπωσδήποτε πρέπει να προβούμε και σε πιλωτικά προγράμματα και ένα σωστό πιλωτικό πρόγραμμα θα ήταν δωρεά πρόσβαση σε Wi-Fi σε μια απομακρυσμένη περιοχή ή δωρεάν πρόσβαση και Wi-Fi στους νέους ανθρώπους. Μπορούμε να το κάνουμε Πιστεύω ότι είμαστε σύμφωνοι και όταν η Επιτροπή έχει και την στήριξη του Ευρωκοινοβουλίου, τα πάντα μπορούν να γίνουν και η Ευρωπαϊκή Ένωση να αρχίσει να παίρνει τον ρόλο και τον χαρακτήρα που οι νέοι άνθρωποι και όλοι εμεί οροματιστήκαμε. Ευχαριστώ. ευχαριστώ. Βέρνερ, Βέρνερ, Ευχαριστώ θερμά, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα αυτή τη δέσμη μέτρων όπως το προτείνεται σε δύο τμήματα να το διαχωρίσουμε ανταγωνιστικότητα και δεύτερον είπαν αρκετά οι συνάδελφοι πρέπει ταχύτερα να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και σε αυτό πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτή την πρωτοβουλία όπως και στο ταχύ διαδίκτυο παντού, παντού και στις περιφέρειες της υπαίθρου όπου δεν υφίσταται. Πρέπει αυτό να μεριμνήσουμε να το κάνουμε. Το άλλο θέμα, ο προλαλής σας το ανέφερε, είναι για τους πολίτες. Wi-Fi for you. Αναφέρατε ένα θέμα στην αρχή, τις κοινωνικο-οικονομικές πτυχές. Θα ήθελα σε αυτό να υπησέθετε, να μας εξηγήσετε τι εννοείτε. Εγώ για τους πολίτες στην Ευρώπη που ε, ε, ενθουσιάζονται με το Interrail στην Ευρώπη 1,5 δις ετήσια θα στήχιζε. Τώρα 120 εκατομμύρια για τρία χρόνια είναι ψίχουλα σίγουρα και γι' αυτό θα ήμουν υπέρ του να διασφαλίσουμε πιο ισορροπη, ισόρροπες σχέσεις το να το διαχωρίσουμε σε τρία σημεία και όταν βλέπουμε ότι ουσιαστικά δεν είναι ισορροπημένες οι σχέσεις αυτές πρέπει κάτι να κάνουμε με αυτά τα κονδύλια μπορούμε να προσπαθήσουμε όμως να δημιουργήσουμε ένα ενθουσιασμό στους πολίτες για την Ευρώπη και να κινητοποιηθούν. Θα πρέπει να βελτιώσουμε λοιπόν τα πράγματα, να είμαστε πιο ισορροπημένοι λοιπόν και να θεσπίσουμε προτεραιότητες, ιδιαίτερα για την μεγαλύτερη εισαγωγή της πέμπτης γενεάς 5G, της πέμπτης γενεάς που είναι πολύ σημαντικό να είμαστε ταχύτεροι ακόμα γι' αυτό. Ευχαριστώ συνάδελφε Βέρνερ. συνάδελφε Κέλλη έχετε το λόγο. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Τα σχόλια έδειξαν ότι υπάρχει ομοφωνία. Είναι πολύ καλό αυτό το αποτέλεσμα σε οποιαδήποτε επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου. Αλλά έχει νόημα να υπάρχει συμφωνία, γιατί αυτό προτείνεται είναι απαραίτητο κυρίως αν θέλουμε να αποκριθούμε στους στόχους που έχουμε θέσει. Δεν θέλουμε να είμαστε οι πλέον ανταγωνιστικοί στον κόσμο και προσπαθώντας να αναζωογονήσουμε κυρίως την Ήπεθρο. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει αν ε, ταχείας ευρυζωνικής και διασυνδέσεων ε, Wi-Fi σε όλη την Ευρώπη. Αυτό πρέπει να κάνουμε θα είναι να καταλήξουμε σε ένα πραγματιστικό σχέδιο και να πούμε σε κάθε περιφέρεια, ανεξάρτητα πόσο θα χρειαστεί μέχρι το 2018-2020 η περιοχή σας θα συνδεθεί κανονικά με όλα τα σύγχρονα μέσα για να μπορεί να κινηθεί στο ψηφιακό κόσμο. Και μετά να πάμε να απευθυνθούμε στα κράτη-μέλη. Κυρίως το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο να πετύχουμε κονδύλι του προπολογισμού για να πετύχουμε αυτό το σκοπό. Τώρα που έφυγε ο Ντέιβιτ Κάμερον, που ήταν υπεύθυνο για τη μείωση του προπολογισμού την προηγούμενη φορά, ίσως να υπάρχει μεγαλύτερος ρεαλισμός σχετικά με το τι μπορεί να πραγματοποιήσει η Ευρώπη με πιο οικονομικό τρόπο στο σύνολό της δηλαδή να κινηθεί η Ευρώπη με καλύτερα αποτελέσματα από ό,τι αν κινηθούν τα κάτι μέλη μεμονωμένα. Αυτό έχω να προτείνω. Δεύτερον, παράδειγμα του τι μπορεί να επιτευχθεί. Στη δική μου εκλογική περιφέρεια, στο West Cork, στο Σκιμπερίν, σε μικρή πόλη, δημιουργήθηκε λοιπόν ένας κόμβος εκεί, με ταχεία ευρυζωνική και διάφορες υπηρεσίες και η πόλη μεταμορφώθηκε. Αν μπορεί αυτό να επαναληφθεί και αλλού, κυρίως η Ήπεθρος θα αναζωογονηθεί. Ευπρόσδεκτες οι προτάσεις σας λοιπόν. Αυτά που είπαν οι συνάδελφοι όσον αφορά τεχνολογία πέμπτης γενιάς είναι σωστά. Είπατε ότι είναι απλώς η κίνηση. Η κίνηση με μίζα ή με μανιβέλα, να ξεκινήσει ο κινητήρας, θέλω να πάρει μπροστά. Λοιπόν, από τη στιγμή που ξεκινήσει ο κινητήρας, θα δημιουργηθεί, θα κινηθούμε, θα δημιουργηθεί ε, αδράνεια κινητική και θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε και μπορούμε να το υποστηρίξουμε σαν εγχείρημα. Ευχαριστώ συνάδελφε Κέλλη. Συνάδελφε Βυρκούνεν, έχετε το λόγο. Κυρία Βυρκούνεν, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρότασή της. Είναι πολύ σημαντικό να προσέξουμε το πώς θα επιταχυνθούν οι επενδύσεις για υποδομές. Η ζήτηση για κινητά δεδομένα αυξάνεται κατά 60 με 100% το χρόνο. Και είναι σίγουρο ότι η σημερινή χωρητικότητα δεν αρκεί για μελλοντικές υπηρεσίες. Δεν υπάρχει μία λύση για όλα τα πράγματα. Χρειαζόμαστε διαφορετικά εργαλεία σε διάφορες ε, περιοχές για να ενθαρρυνθούν οι επενδύσεις. Άρα είναι σημαντικό να εστιαστούμε επί των υποδομών τώρα, διότι πρέπει να επιταχυνθούν οι διασυνδέσεις σε όλη την Ευρώπη, σε όλες τις περιοχές. Τώρα αναφερόμενοι στην ασφάλεια. Θα πρέπει οι καταναλωτές να κινούνται σε ένα ασφαλές περιβάλλον, ψηφιακό. Πρέπει να προσέξουμε όμως να μην ρυθμίσουμε υπερβολικά τον τομέα της πληροφορικής. Η Ευρώπη πρέπει να βρει σωστή ισορροπία στην προσέγγιση μεταξύ ασφαλείας και ανοιχτής προσέγγισης, μεταξύ νομοθεσίας και ευελιξίας. Διότι ελευθερία και ασφάλεια δεν είναι αλληλοσυγκριόμενες έννοιες, μπορούν να προωθήσουν τον ίδιο στόχο να οδηγηθούμε στην ψηφιοποίηση των υπηρεσιών και της βιομηχανίας. Αν θέλουμε να έχουμε θέσεις απασχόλησης και ανάπτυξη στην Ευρώπη και ανοιχτό ψηφιακό κόσμο για όλους στην Ευρώπη, θα πρέπει να είναι ανοιχτή η Ευρώπη για τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα που επιφέρει η ψηφιοποίηση για να είμαστε ανταγωνιστικοί και να ανταποκριθούμε στην ταχύτητα των εξελίξεων τα ανοιχτά, ε, τα ανοιχτά προγράμματα οδήγησαν σε καινοτομίε και σε νέα επιχειρηματικά μοντέλα. Θα πρέπει να είναι ανοιχτά ε, τα προγράμματα για να προωθηθούν νέε ιδέε, να είναι ε, πιο ελεύθερη η διάθεση των στοιχείων. Θέλουμε λοιπόν να γίνουν επενδύσεις, να αυξηθεί η διασυνδυσιμότητα στην Ευρώπη, να έχουμε ένα ασφαλές περιβάλλον για όλους στον ψηφιακό κόσμο. Για να τα κάνουμε αυτά πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, να μην προσπαθήσουμε να ρυθμίσουμε τα πάντα στον τομέα της ψηφιακής ε, τεχνολογίας και της πληροφορικής. Ευχαριστώ, ολοκληρώθηκαν οι παρεμβάσεις. Ήμασταν πάρα πολύ καλοί με το χρόνο, πολύ πειθαρχημένοι. Έχουμε, θα έλεγα, και ένα πεντάλεπτο ό,τι χρειάζεται για να δώσετε τις απαντήσεις σας. Δεν θα ήθελα να σας περιορίσω χρονικά για να μπορέσετε να καλύψετε τις ε, ερωτήσεις που ετέθησαν. Ευχαριστώ. Εφόσον δεν έχουμε πολύ χρόνο, θα εστιαστώ επί των βασικών σημείων που ακούστηκαν και νομίζω τέσσερα ακούστηκαν. Ήταν τέσσερα. Ευχαριστώ όμως όλους και ευχαριστώ και την κυρία Δεκαστήλιο για την στεναρή αυτή παρέμβασή της. Εσείς αναφέρατε ένα θέμα για την Κοινοβουλευτική Επιτροπή και το Κοινοβούλιο γενικά για το κόστος αυτό το οποίο θα συνεπάγεται. Ο Αντιπρόεδρος όταν είχε προσέλθει, φυσικά από πλευρά της Επιτροπής αναγνωρίζουμε για την εσωτερική αγορά για το κόστος και για το, τους, το κωδικό αναχώρα και το κόστος Πιστεύουμε ότι το πακέτο αυτό τώρα με την πίεση την ανταγωνιστική που θα δημιουργήσει και που θα δημιουργήσει πολλές δυνατότητες υπάρχει ένα στοιχείο για την αντιμετώπιση των ρητρών εκπνοής, ε, λήξης ε, συμβάσεων και συμβολέων. Αυτό θα κάνει και διαφορά. Δεν υποεκτιμούμε όμως ε, και την πολιτική εμβέλεια αυτών των σημείων. Τώρα, μερικές πτυχές ένα θέμα για τις προτεραιότητες που είπατε ότι μπορεί να είναι πιο φιλόδοξες Άλλος ρώτησε ποιες είναι οι προτεραιότητες. Για μερικά παραδείγματα σε σχέση με το θέμα των επενδύσεων που έχει τεράστια σημασία και το θέμα του φάσματος που είναι σπουδαίας ε, ε, έχει και αυτό τη σπουδαιότητά του. Αν δούμε λοιπόν όλο το πακέτο δεν είναι μόνο το νομοθετικό τμήμα και ε, οι διατάξεις ε, είναι το να υπάρξει πίεση να μπορέσουν όλα έγκαιρα να λειτουργήσουν και γοργά κάνουμε λόγο για πράγματα τα οποία δεν χρειάζονται νομοθεσία για να λειτουργήσουν. Με τα σωστά λοιπόν μηνύματα που μπορούν να επεμφθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μπορούμε να δράσουμε ταχύτερα. Τώρα, τι θα γίνει με τις δημόσιες επενδύσεις, ιδιωτικές επενδύσεις, υπολογίζονται τεράστιες επενδύσεις που θα είναι αναγκαίες ε, για αυτόν τον τομέα και τα δημόσια κονδύλια. Είπε ο κύριος Κέλλη ότι χρειάζονται περισσότερα, περισσότερα για την ε, ε, προσπάθεια αυτή, αλλά στο τέλος τέλος πρέπει να μπορέσουν να συνδυαστούν και τα κρατικά, τα δημόσια κονδύλια και οι ιδιωτικές επενδύσεις. Πρέπει να δημιουργηθεί το σωστό πλαίσιο ώστε να μπορέσει αυτό να λειτουργήσει στο συνδυασμό αυτό σωστά. Για την πέμπτη γενεά ε, με χαρά βλέπουμε ότι υπάρχουν, ε, υπάρχει ενδιαφέρον και υπάρχουν και νέες ιδέες πώς μπορεί να προχωρήσει αυτό. Βρισκόμαστε στη σωστή πορεία. Αν, μπορούμε να μπορέσουμε, αν μπορέσουμε να λειτουργήσουμε έτσι ευθύς εξ αρχής, ίσως θα μπορέσουν αυτά να καλυφθούν στη συνέχεια. Και για να είμαστε συνεπείς, φυσικά πρέπει να είμαστε συνεπείς για αυτό το οποίο κάνουμε και πώς αντιμετωπίζονται τα κράτη-μέλη και πώς θα μπορέσουμε να κινηθούμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Αυτά είχα να πω και κάλυψα νομίζω αυτά που χρειαζόντουσαν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Εκτιμήσαμε τη σαφήνειά σας. Είμαι σίγουρη ότι έχουμε δυνατότητα σύντομα να συναντηθούμε και να συζητήσουμε τα θέματα. Στο επανειδήν. Θα αλλάξουμε τώρα θέμα για μια στιγμή. No, no, yo no, el primo, el Λοιπόν, συνεχίζουμε τις εργασίες μας. Το δεύτερο θέμα στην ημερησία διάταξη έχει μεγάλη σημασία και συνδέεται με το προηγούμενο είναι η έκθεση για την ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Θα δώσω αμέσως το λόγο στον συνάδελφο Beauty Coffer. Thank you. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ Πρόεδρε, συνάδελφοι. Πραγματικά πρέπει να πω ότι πιστεύω ότι δύσκολα μπορεί να υπερεκτιμήσει κανείς ε, τη σπουδαιότητα αυτού του θέματος για το μέλλον της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και ιδιαίτερα επίσης για το μέλλον της ευρωπαϊκής ε, παραγωγής. Προτού όμως ε, κάνω κάποιες παρατηρήσεις σε σχέση με την ουσία του θέματος, κάποιες διαδικαστικές δηλώσεις τοποθετήσεις. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, όπως έχει σχεδιαστεί, το σχέδιο έκθεσης θα περάσει προς μετάφραση αρχές Δεκεμβρίου και η εξέταση του σχεδίου έκθεσης προβλέπεται για ε, νωρίς το Γενάρη, τον Ιανουάριο, 12 Ιανουαρίου συγκεκριμένα. Θα ψηφίσουμε σε αυτή την Κοινοβουλευτική Επιτροπή το Μάρτιο θα ψηφίσουμε στην Ολομέλεια πιθανότατα τον Απρίλιο. Πέρα από αυτά, διαδικαστικά, θα έπρεπε να αναφέρω ίσως ότι η Επιτροπή Ίνκο και η Επιτροπή Κάρτ Πολιτισμού έχουν <clears throat> σε σχέση με το, το άρθρο 50 συν ε, το καθεστώς το οποίο έχουν για ε, να μπορούν να συμπεριληφθούν και συμμετάσχουν με τις, ε, τα προνόμια και τα δικαιώματα αυτά σε αυτές τις εργασίες μας. Όπως είπα, σε σχέση με αυτές τις παρατηρήσεις, η επόμενη φάση για την παραγωγή είναι ο οποιοδήποτε που μπορεί να ε, παίξει και να συμμετάσχει. Όλα όμως εξαρτώνται από το πώς εμείς θα διαχειριστούμε τη μεταβατική περίοδο προς την ε, ψηφιοποιημένη βιομηχανία. Η Ευρώπη έχει, και το πιστεύω αυτό στεναρά, πολύ καλές προϋποθέσεις, θετικότατους όρους και προϋποθέσεις, πολύ μεγάλο δυναμικό, αλλά θα μπορέσουμε μόνο να πετύχουμε σε αυτό το εγχείρημα, σε αυτόν τον αγώνα δρόμου, ώστε να είμαστε ηγέτες, να έχουμε ηγετικό ρόλο και να μπορέσει να μεταμορφωθεί η οικονομία μας με επιτυχία αν δράσουμε στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, στην ευρωπαϊκή σκηνή, ενιαία. Ακούσατε όλοι να επαναλαμβάνει αυτό το μήνυμα μέχρι κορεσμού ε, μέχρι ε, εξάντλησης ε, και αν δεν υπάρξει μια συντονισμένη ευρωπαϊκή στρατηγική δεν θα τα καταφέρουμε. Και επίσης θα ήθελα με αυτή την ευκαιρία να αναφέρω ότι πιστεύω εγώ προσωπικά ότι πρόκειται για μια εγκάσια ως θέμα ύλη που καλύπτει πάρα πολλά διαφορετικά πεδία και τομείς πολιτικής και διαμόρφωσης πολιτικής. Π.χ. για παράδειγμα πώς θα αντιμετωπίσουμε το θέμα του FDI υπό το πρίσμα της ψηφιοποίησης είναι ένα από αυτά. Όπως τονίστηκε πρόσφατα στη ε, δημόσια στη Γερμανία με την εξαγορά εν, ενός από ε, ε, των κοσμημάτων ε, την εταιρεία Κούκα από μια κινέζικη εταιρεία στο Guangdong βλέπουμε ότι αυτή είναι ακριβώς μια πτυχή που πρέπει να λάβουμε οπωσδήποτε υπόψη τι γίνεται και τι τεκταίνεται σε αυτόν τον τομέα. Ψηφιοποίηση. Πρόκειται φυσικά για τεχνολογία, αλλά και για κάτι παραπάνω από την τεχνολογία. Πρόκειται για την ανάπτυξη τεχνολογίας με μεγατάσεις, με την παγκοσμιοποίηση και ε, ε, θέματα που πρέπει να ε, μας ευαισθητοποιήσουν σε παγκόσμια κλίμακα. Να δημιουργηθεί λοιπόν μια σωστή βάση για τις ευρωπαϊκές προσπάθειες. Αν τα καταφέρναμε να διασυνδέσουμε την ψηφιοποίηση, τα στοιχεία για την ψηφιοποίηση μέσα στο πλαίσιο πολιτικής καινοτομίας από πλευράς έρευνας και της αηφορίας αυτής της στρατηγικής καινοτομιών. Επιτρέψτε μου να αναφέρω κάπως πιο εξειδικευμένα σημεία, δεν θα μακρηγορήσω νομίζω ότι θα πρέπει να εξετάσουμε και την χρηματοδότηση, τα κονδύλια που θα διαθέσουμε. Θα πρέπει επίσης να εξετάσουμε πιο εξειδικευμένα και για το πώς θα συμμετέχουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε αυτό το πλαίσιο, ποιος θα είναι ο ρόλος τους και ποιες επιδόσεις πρέπει να έχουν διότι θα λέγαμε και θα συμφωνούσατε σίγουρα μαζί μου ότι αν δεν συμπεριληφθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι ΜΜΕ, σε αυτή τη στρατηγική ψηφιοποίηση από πλευράς της Ευρώπης, δεν θα μπορούσαμε να πετύχουμε, να καταφέρουμε, να επιτύχουμε τους στόχους μας. Και να δούμε επίσης και τι κάνουν και οι ανταγωνιστές μας σε αυτούς τους τομείς. Ίσως θα μπορούσαμε κάποια μαθήματα να συναγάγουμε, ώστε να μπορέσουμε να είμαστε πιο επιτυχείς ίσως. Σίγουρα πρέπει να δούμε και τις υποδομές. Δεν μακρηγορεί κανείς λέγοντας το αυτό. Πρέπει να, και η τυποποίηση να συμπεριληφθεί, standardization, που ε, υπάρχει για την ψηφιοποίηση και ζήτημα σε σχέση με την τυποποίηση. Έχουμε και την εκμετάλλευση του ανθρώπινου δυναμικού που έχουμε στη διάθεσή μας και αυτό πρέπει να λάβουμε υπόψη και σίγουρα να μην αμελήσουμε, να μην ξεχάσουμε και την προστασία ε, σε σχέση με ε, τα θέματα και των εργαζομένων και των ε, δεδομένων όσον αφορά την ε, δημιουργία ενός ε, νέου πλαισίου ψηφιοποίησης στο βιομηχανοποιημένο κόσμο. Έχω επαφές με τους σκιώδεις εισηγητές, ευελπιστώ ότι θα βρούμε κοινά στοιχεία και προσβλέπω σε μια γόνιμη διαδικασία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον συνάδελφο Μπουτικόφε ο οποίος σίγουρα θα κάνει μια εξαιρετική δουλειά. Θα ήθελα και εγώ να κάνω μια παρατήρηση σαν σκιώδης εισηγήτρια των σοσιαλιστών, όπως είπε και ο Μπούτι Κόφερ, νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία για να μην πω μια απέτηση για μας, το να προσπαθήσουμε να προσαρμόσουμε το παραγωγικό δυναμικό της υπήρου μας σε επίπεδο ε, αηφορίας και σε σχέση βέβαια με αυτά τα οποία γίνονται στον υπόλοιπο κόσμο. Έχουμε βέβαια κάποιες δυσκολίες τις οποίες ανάφερε ήδη ο κύριος ε, ε, Beauty Coffer. Η πραγματικότητα των καινοτομιών στην Ευρώπη βρίσκεται σε διαφορετικά επίπεδα. Υπάρχουν πολύ σημαντικές διαφορές ανάμεσα σε χώρες, σε κάποιες υπάρχουν διαμάντια παραγωγικά. Υπάρχουν όμως και κάποιες μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ψηφιοποιηθεί σε ελάχιστο επίπεδο δυστυχώς όν δει κανεί πόσες ευρωπαϊκέ επιχειρήσεις χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για τις εμπορικές τους δραστηριότητες, εκπλήσεται από το χαμηλό ακριβώ επίπεδο. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια προσπάθεια προσαρμογής και θα πρέπει ε, να συμμετέχουν ακόμα και οι μικρομεσαίες οι οποίες ε, δεν έχουν καταφέρει να συνδεθούν μεταξύ τους. Πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να πετύχουμε τους στόχους μας όχι μόνο με κάποιους πρωταθλητές μεμονωμένους <clears throat> αλλά συνδυάζοντας ε, τις παραγωγικές δυνατότητες όλων των τεχνολογικών τομέων. Να υπάρξει μια διάδοση δηλαδή των σημαντικών αυτών βημάτων που πρέπει να γίνουν και σε επίπεδο υποδομών και σε επίπεδο γενικά αρμοδιοτήτων και γνώσεων μια σειρά από δραστηριότητες οι οποίες θα μπορέσουν να λάβουν υπόψη τους την ανάγκη για ψηφιοποίηση. Εκεί λοιπόν υπάρχουν σημαντικές δυσκολίες. Σε κάποια κρατημέλη είπαμε τα πράγματα έχουν κάπως προχωρήσει έχουν υπάρξει κάποια βήματα προόδου. Από την άλλη σε άλλες χώρες δεν έχει υπάρξει η απαιτούμενη επεξεργασία μιας κάποιας στρατηγικής. Νομίζω λοιπόν ότι η παρέμβαση η οποία πρέπει να γίνει είναι μια ευκαιρία έτσι ώστε να υπάρξει αναγνώριση της πραγματικότητας που ισχύει σε κάθε χώρα για να μπορέσουμε εμείς να ξεπεράσουμε αυτή την έλλειψη ισορροπίας η οποία καθίσταται σταδιακά σαν στοιχείο αποδυνάμωσης του συνόλου του παραγωγικού μας δυναμικού. Πρέπει να θέσουμε λοιπόν το πρόβλημα και σε σχέση με τη δημιουργία θέσεως, θέσεων απασχόλησης, γιατί το ίντερνετ των πραγμάτων θα αλλάξει την πραγματικότητα των γνώσεων, της εργασίας και την ίδια την έννοια της απασχόλησης θα έλεγα. Εγώ βλέπω στη χώρα μου σαν παράδειγμα κάποιες μελέτες οι οποίες προωθούνται από τους συνδικαλιστικούς κύκλους που προσπαθούν να δουν τι πρέπει να γίνει και τι μπορούν να κάνουν. Αλλάζοντας το ίδιο το προφίλ της βιομηχανικής πραγματικότητας στην Ευρώπη, ε, θα πρέπει να δούμε ακριβώς τι ρόλος επιφυλάσσεται για το ανθρώπινο δυναμικό, για τον ανθρώπινο παράγοντα. Είναι βασικό λοιπόν να προχωρήσουμε σε αυτό το μήνυμα. Λοιπόν, εγώ σαν σκιώδης θα συνεργαστώ με τον εισηγητή. Το σύνολο γενικά της πολιτικής μου ομάδας θέλει να βοηθήσει. Α, συγγνώμη, ε, ξέχασα την πρώτη στη σειρά, την κυρία Καστίγιο. Νόμιζα ότι θα μιλούσατε στον επόμενο γύρο σας. Δίνω αμέσως το λόγο, κυρία Καστίγιο. Ευχαριστώ από πλευρά ε, του συναδέλφου που είναι σκιώδης εισηγητής για μα. Ε, για τι εξής ιδέε. Πρώτον, οι παραγωγοί θα επιβιώσουν μόνο αν θα μπορέσουν ε, να ανέβουν στο τρένο της ψηφιακής οικονομίας. Θα πρέπει οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να υποφεληθούν. Υπάρχουν περιορισμένες δυνατότητες και θα πρέπει να ευχηθούμε να μπορέσει κάθε επιχείρηση να συμμετάσχει πλήρως ε, σε αυτό το εγχείρημα, άσχετα ποιες είναι οι διαστάσεις της. Υπάρχει η ανάγκη να μην υπάρχουν υπερβολικές ε, ρυθμιστικές επιβαρύνσεις για να προαχθεί και να μην υπάρξουν προσκόμματα για την καινοτομία και για την εθνική, τις εθνικές πρωτοβουλίες ε, μέσα σε ένα ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να προχωρήσουμε για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε περισσότερες επενδύσεις και να μπορέσουν να προαχθούν οι δυνατότητες για την ψηφιοποίηση. Η τυποποίηση όπως αναφέρθηκε, η διαλειτουργικότητα των συστημάτων και ούτω καθεξής είναι σημαντικές υποθέσεις. Η εμπιστοσύνη είναι σημαντική υπόθεση και αυτή. Θα πρέπει να δοθούν κίνητρα για να υπάρξει καινοτομία. Ταυτόχρονα θα πρέπει από πλευράς των δυνατοτήτων να μπορέσουν να υποφεληθούν ε, πολλαπλά όλοι οι εμπλεκόμενοι. Εδώ θα πρέπει να βρεθεί η σωστή ισορροπία σε σχέση με την προστασία και την εμπιστοσύνη και την διευκόλυνση που θα πρέπει να ε, διασφαλίζεται για τις επιχειρήσεις στην αγορά. Να, αν δεν δημιουργηθεί ένα δίκαιο πλαίσιο στην αγορά δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε το δίκαιο θα πρέπει να σχεδιαστεί ώστε να μπορέσουν να, να ρυθμιστούν οι εκκρεμότητες ώστε να είναι πλήρως δίκαιο το πεδίο δραστηριοποίησης για την καινοτομία. Πρέπει να εξεταστεί επίσης ε, η προαγωγή των σωστών προδιαγραφών ώστε να μπορέσουμε στην, στο θεματολόγιο να δράσουμε αποτελεσματικά και τέλος θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η ανάγκη να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης ε, σε, στην ψηφιακή οικονομία μέσω της προσπάθειας μας αυτής. Ε, σας ευχαριστώ πολύ. Αυτές είναι οι απόψεις του συναδέφου που απουσιάζει. Ευχαριστώ Πιλάρ. Δεν έχω δει ποτέ το Σαλίνι, με ξανθό μαλλί, μπερδεύτηκα. Σας ευχαριστώ. ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ναι, τον εισηγητή. Έχουμε ήδη συναντήθει και πραγματικά εκτίμησα και εκτιμώ την προσέγγιση για αυτό το θέμα. Η ψηφιοποίηση είναι ένα ευρύτατο θέμα και καλύπτει όλες τις άλλες πολυσχηδείς πτυχές, βιομηχανικές πτυχές και ζητήματα όπως επίσης και το επιχειρήν από πλευρά των επιχειρήσεων στην Ευρώπη. Αντιμετωπίζουμε τεράστιες προκλήσεις στην Ευρώπη, τεράστιες αλλαγές και μεταβολές και θα πρέπει να παρκέσουμε, να βρούμε την πιο αποτελεσματική όδο για να διασφαλίσουμε την ανταγωνιστικότητά μας και τα συμφέροντά μας και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι αυτά όλα θα αποφασίσουν, θα είναι αποφασιστική σημασία για τις επιχειρήσεις και παγκόσμια. Συμφωνώ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι οι βιομηχανίες, οι επιχειρήσεις ε, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα και να υποφεληθούν από την ψηφιοποίηση. Και θα πρέπει να διευκολύνουμε ε, τις δυνατότητες ώστε να υπάρξει επαρκής χώρος να δράσουν σε ένα διεθνές πλαίσιο με τα ε, μέγα δεδομένα, με, τις, ε, με τη ρομποτική, με τις ε, νεότερες τεχνολογίες. Το σημαντικό είναι ότι ίσως θα πρέπει να αφουγκραστούμε και να δούμε τι συμβαίνει και στις συναντήσεις της ΣΤΟΑ για την, ε, τα θέματα τεχνολογίας, ενοτομίας και έρευνας και σε σχέση με την διαμόρφωση της αγοράς εργασίας, ε, του πλαισίου ε, θα έλεγα, του περιβάλλοντος του εργασιακού που με τις αλλαγές και τις μεταβολές υπάρχουν επιπτώσεις σε όλη την Ευρώπη. Αυτά μπορεί να δημιουργήσουν και πραγματικά πολύ μεγάλη μεγάλη εντύπωση, ίσως και φόβο. Είναι τεραστίων διαστάσεων. Συμφωνώ λοιπόν με τον εισηγητή ότι ουσιαστικά πρέπει σίγουρα να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει διασύνδεση μεταξύ της παιδείας, εκπαίδευσης, κατάρτισης όλων των τομέων με αυτή την προσπάθεια. Θα υπάρξουν ευρύτατες αλλαγές, θα υπάρξει πίεση και ε, απαιτήσει, ε, ζήτηση για δεξιότητες, ικανότητες, ε, όλα αυτά θα διαμορφώσουν το μέλλον μας. Θα εξαρτηθεί από την ετοιμότητα και προθυμία μας να συμπορευτούμε. Γι' αυτό είναι σημαντικότατο να συνοδεύσουμε την ψηφιακή καινοτομία με τις αναγκαίες επενδύσεις. Επίσης αυτά πρέπει να ληφθούν ιδιαίτερα υπόψη όταν κάνουμε λόγο για σημαντικές πρωτοβουλίες όπως τον ορίζοντα 2020, Horizon 2020, να διευκολύνουμε τα μέσα και τις δυνατότητες να προχωρήσουμε. Συμπεραίνω, ευχαριστώ τον εισηγητή και προσβλέπω στη μελλοντική μας συνεργασία. Και πιστεύω πράγματι ότι τα καλύτερα ε, στοιχεία είναι τα μηνύματα που στέλνουμε για αυτούς τους τομείς. Θα πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας να εμπλακούμε σε αυτή την προσπάθεια και ευελπιστώ ότι θα, καταφέρουμε, θα τα καταφέρουμε αν προσπαθήσουμε από κοινού. Ευχαριστώ. <coughs> Ευχαριστώ. Συνάδελφε Νόχαουζεν, ελπίζω να μην σκότωσα το όνομα σας. Πολύ καλά, Κύριε Νόχαουζεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συμφωνώ με τα περισσότερα από αυτά που είπαν οι συνάδελφοι. Ο κ. Μπίτεχόφερ το είπε σωστά. Δεν πρέπει να υποτιμούμε αυτά που συμβαίνουν όσον αφορά τον ψηφιακό κόσμο και την ψηφιοποίηση της οικονομίας, όχι μόνο της βιομηχανίας. Δεν ζούμε σε εποχή αλλαγών, αλλά σε αλλαγή εποχής, άμα μιλάμε για την ψηφιοποίηση. Πότε ήταν τελευταία φορά που χρησιμοποίησαμε ε, τηλεφωνικό κατάλογο από χαρτί. Χτες που έκλεινα ξενοδοχείο μέσω του booking.com σκεφτόμουν αυτή τη συζήτηση και έλεγα σχεδόν πρόσφατα έπρεπε να τηλεφωνάμε στα ξενοδοχεία για να κλείσουμε και να βρούμε ξενοδοχείο. Άλλαξε η ζωή μας τόσο πολύ και όταν περπατάμε στο δρόμο για να πάμε στο ξενοδοχείο Μπορούμε να ζητήσουμε, αν δεν θέλουμε να περπατήσουμε, να καλέσουμε ταξί από το Uber και να μην ψάχνουμε να βρούμε πού κάνουν στάση τα που έχουν, ε, περιμένουν, έχουν πιάτσα τα ταξί. Λοιπόν, είδαμε τις αλλαγές που συμβαίνουν και στη βιομηχανία. Έχει πολλά να κερδίσει η βιομηχανία από την ψηφιοποίηση. Όπως ανέφεραν συνάδελφοι, είναι το διαδίκτυο των πραγμάτων, είναι τη διάστατη εκτύπωση, τα big data, τεχνητή νοημοσύνη, η ρομποτική, όλα αυτά συμβαίνουν ταυτόχρονα. Θα πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Η ζωή για του εργαζομένους θα γίνει ασφαλέστερη, διότι μπορούν τα ρομπότ να λάβουν επικίνδυνη εργασία, την καταπολέμηση των πυρκαγιών, ή για την αφαίρεση αμοιάντου μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τεχνολογία για βελτιώσεις. Απ' την άλλη συμφωνώ με αυτά που είπαν οι συνάδελφοι ότι κάποιες από τις νέες θέσεις εργασίας απαιτούν νέες δεξιότητες, νέου τύπου εκπαίδευση και θα πρέπει το εργατικό δυναμικό να αντέχει στις αλλαγές. Όλοι θα πρέπει να μπορούν να συμμετέχουν στη νέα οικονομία με νέες δεξιότητες. Οπότε ένα θεματολόγιο με νέε δεξιότητε είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι τη όλη προσπάθεια. Σαν δημόσιο τομέα πρέπει να εστιαζόμεθα όχι μόνο επί τη παιδεία, αλλά και επί άλλων προποθέσεων που χρειάζεται βιομηχανία. Για να είναι ανταγωνιστική στο παγκόσμιο προσκήνιο. Χρειαζόμαστε τη διασυνδεσιμότητα, κάτι που αναφέρθηκε στην πρώτερη συζήτηση. Δεν θα επαναλάβω τα υποθέντα. Κάτι που δεν αναφέρθηκε είναι η κβαντική υπολογιστική. Έχουμε 7,5 δισεκατομμύρια ανθρώπους που συνδέονται μεταξύ τους. Αλλά ήδη τώρα έχουμε 22 δισεκατομμύρια συσκευές συνδεδεμένες με το διαδίκτυο των πραγμάτων, των αντικειμένων. Έχουμε εκθετική ανάπτυξη εκεί. για να χρησιμοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες χρειαζόμαστε πάρα πολύ μεγάλες υπολογιστικές δυνατότητες και μόνο με την κβαντομηχανική και την κβαντική υπολογιστική μπορούμε να τα πετύχουμε. Βλέπω να βοσβήνει το φως, έχω περάσει το κόκκινο, τελείωσε ο χρόνος μου. Αυτά ίσως τα πω την επόμενη φορά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και για αυτή τη, αυτά που μας είπατε. Συνάδελφα την πρόεδρε Κόλιτσεκ, έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Έχω προσωπική εμπειρία αυτών. Ξέρω κάτι από τον αυτοματισμό στη βιομηχανία και τη σχετική νομοθεσία. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα για την παραδοσιακή βιομηχανία ήταν η μετακίνηση από αναλογικές ε, μηχανές και μηχανήματα και συσκευές προς ψηφιακές. Η ψηφιοποίηση των σημάτων ήταν ένα πρόβλημα που χρειάζεται για να λειτουργήσει η βιομηχανία. Η ψηφιοποίηση μας επιτρέπει ε, να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Ε, αυτό που μας παρουσίασε πολύ ωραία στην εισαγωγή του ο κύριος συζητητής. άλλη η προσέγγιση των ανθρώπων στις αναλογικές συσκευές από τις ψηφιακές. Ποια είναι η σχέση όμως των ανθρώπων με τη δημόσια διοίκηση και με την τοπική αυτοδιοίκηση. Ε, οργάνωση, μεταφορές, τελικά προϊόντα, ε, όλα αυτά επηρεάζονται από την ψηφιακή τεχνολογία και τα δίκτυα, είτε είναι μεταφορικά δίκτυα, είτε είναι οδικά δίκτυα. Τα δίκτυα παίζουν σημαντικό ρόλο. Και η δημόσια διοίκηση και η τοπική αυτοδιοίκηση, οι δήμοι και οι κοινότητε κερδίζουν από τη συλλογή στοιχείων. Για να πετύχουν τη συλλογή των στοιχείων χρειαζόμαστε κοινά πρότυπα, συμπεφωνημένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την ανταλλαγή στοιχείων. Αυτό δεν είναι μόνο σημαντικό για τη βιομηχανία και άλλου τομεί. για τη δημόσια διοίκηση, για, την, ε, για τους δήμους, της κοινότητας, την τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι σημαντικά αυτά. Χρειάζονται δεδομένα τα οποία ε, συμμορφώνονται με κοινέ προδιαγραφές για να γίνεται σωστή η χρήση τους. Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι δεν πρέπει να προσέξουμε μόνο πώς θα εκπαιδευτούν οι μελλοντικέ γενιές, αλλά και με τους τωρινούς ανθρώπους και εργαζομένους. Τι θα κάνουμε. Εγώ ήμουνα δραστήριο στα τελευταία χρόνια. Αν ήμουν στι μεταφορές και θέλω να ξαναγυρίσω σε, εργο... σε εργοστάσιο παραγωγής γυαλιού, όπως ήμουνα παλιά, πρέπει να, τώρα να προσαρμοστώ και να μάθω πολλά καινούργια πράγματα. Παρόλο που έκανα αυτή τη δουλειά στο παρελθόν. Θα με βοηθούσε η εκπαίδευσή μου και η εμπειρία μου να α, χωνέψω τις νέες γνώσεις. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, 50 χρονών, τόσο στην ηλικία μου, για τους οποίους θα ήταν πιο δύσκολο κάτι τέτοιο. Όταν μιλάμε για ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής οικονομίας, να μην ξεχνάμε και τους ανθρώπους που είναι 50 ετών και άνω. Ε, είναι πολύ σημαντικό, είναι μεγάλο κομμάτι του εργατικού δυναμικού αυτοί οι άνθρωποι. Πρέπει να τους λάβουμε υπόψη. Και αν δεν τους εκπαιδεύσουμε σωστά να προσαρμοστούν, αν δεν τους βοηθήσουμε, προφανώς οι περαιτέρω εξελίξεις θα εμποδιστούν, κυρίως για τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις όταν μιλάμε για την ψηφιοποίηση και την εφαρμογή της ψηφιοποίησεως. Δεν θα γινόταν σε επαρκές βάθος η ψηφιοποίηση, αν δεν το προσέξουμε αυτό. Για να αποκομίσουμε όλα τα αγαθά της ψηφιοποίησης, χρειάζεται εις βάθος προσέγγιση για να δρέψουμε τους καρπούς της ψηφιοποίησης. Πρέπει όλοι οι άνθρωποι που κινούνται σε αυτόν τον τομέα, στον παραγωγικό, να καλυφθούν και να εκπαιδευτούν. Μην ξεχνούμε αυτή την κοινωνική πτυχή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ο κύριος Ταμπουράνο έχει το λόγο. Πράγματι έχουν προχωρήσει οι τεχνικές και στα πλαίσια του βιομηχανικού σχεδίου και πραγματικά έχουμε περάσει τώρα στην επόμενη φάση από την τρίτη βιομηχανική επανάσταση. Γνωρίζουμε όμως ότι σε ορισμένες περιοχές του κόσμου το μέλλον είναι ήδη το παρόν. Αντίθετα από την Ευρώπη υπάρχουν περιοχές οι οποίες είναι οργανωμένες και παράγουν με πολύ γρήγορο ρυθμό τέτοιου είδους προϊόντα. Πρέπει λοιπόν να προβλεφθεί μια κατάλληλη εκπαίδευση για τις νέες γενιές. Ε, ήδη ε, CAD e Σε πολλές ε, περιοχές του κόσμου μαθαίνουν ας πούμε την ευκλήδιο γεωμετρία με την βοήθεια του Computer Assisted Design. ενώ εμείς έχουμε απομονωθεί, βρισκόμαστε πίσω και στον τομέα της ρομποτικής θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε επίσης τι γίνεται και με τα προβλήματα που δημιουργούνται στον τομέα της τεχνολογικής ανεργίας και πώς μπορεί να θίξει τους εργαζομένους στον τομέα αυτό. Οι βιομηχανικές επαναστάσεις ναι μεν δημιουργούν και νέες θέσεις ε, εργασίας, αλλά η ρομποτική σαν παράδειγμα δεν δημιουργεί τόσες για να αντισταθμίσει όσες χάνονται. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να αναμένουμε σημαντικές συνέπειες σε κοινωνικό επίπεδο. Πάντα στον τομέα της κατάρτισης είναι το θέμα της μετακίνησης των επιχειρήσεων. Το ίντερνετ των πραγμάτων και τα λοιπά είναι μια μεγάλη ευκαιρία να μετακινηθεί ένα κομμάτι του βιομηχανικού παραγωγικού ιστού της Ευρώπης σε διαφορετικές περιοχές. Ε, πρέπει όμως εμείς να συμβαδίζουμε με τις εποχές, να έχουμε τη σωστή κατάρτιση, γιατί τότε θα υπάρξει μετακίνηση όχι των μονάδων παραγωγής, αλλά των εγκεφάλων. Στην Ιταλία είναι μία από τις χώρες ε, όπου εξάγονται σε εισαγωγικά πάρα πολλοί ε, επιστήμονες που δεν ζουν πια στην Ιταλία, δεν παράγουν στην Ιταλία. Λοιπόν, η ρομποτική και το ίντερνετ των πραγμάτων είναι μια νέα εποχή για την ανθρωπότητα. Ε, νομίζω ότι και θα πρέπει να απελευθερωθούμε από τη σκλαβιά της εργασίας για κάποιο τμήμα της ανθρωπότητας. Θα ήθελα αυτό το νέο πέρασμα να δώσει μια νέα ευκαιρία ε, στον άνθρωπο να γίνει πιο δημιουργικός και να εργάζεται με πιο εφάνταστο τρόπο από ότι ε, το έκανε στο παρελθόν με τρόπο επαναληπτικό και μονότονο. Τα παραγωγικά μας συστήματα τα οποία εξαρτώνται από την μικροηλεκτρονική εξαρτώνται επίσης και από την εξαγωγική τους δραστηριότητα. Θα έχουμε πολλά να πούμε σε αυτό στο μέλλον. Ευχαριστώ κύριε Ταμπουράνο και κύριε Καπέλο. Ευχαριστώ. Με αυτή την ευκαιρία θα ήθελα να πω ότι ο Σκιώδης εισηγητρία για την ομάδα μας για την έκθεση που θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική δηλαδή για τη βιομηχανία και πόσο σημαντικό είναι τα συστήματα αυτά και από την τελευταία λέσχη των 20 G20 που είπαν ότι ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να στρέψουμε μελλοντικά στην ψηφιοποίηση της οικονομίας και των επιχειρήσεων σε παγκόσμια κλίμακα. Και σε αυτό στην έκθεση που εκπονούμε στο Ευρωκοινοβούλιο είναι ένα σημαντικό βήμα διότι για τη βιομηχανία που είναι ο κινητήρας της ε, ανάπτυξης που δεν μπορούμε να απεμπολίσουμε όχι όμως μόνο η ψηφιοποίηση των βιομηχανιών και επιχειρήσεων, αλλά και η ψηφιοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Έχουμε μελέτες που δείχνουν ότι για την, ε, τις επιχειρήσεις αλλά και για την μικρομεσαία, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σημαντική αύξηση παραγωγικότητας μπορεί να επιτευχθεί και πολύ μεγαλύτερη απόδοση κεφαλαίων. Ο Ρόλαντ Μπέργκερ σε μια ευρύτατη μελέτη το κάλυψε αυτό από την οποία μελέτη απορρέει ότι σε σχέση με τις επιχειρήσεις κατά 25% μπορεί να επιτευχθεί αύξηση ακόμα και μεγαλύτερη από 25% αν, υπάρξει, ή αν υπάρξουν οι όροι και οι προϋποθέσεις ώστε να προχωρήσουμε σωστά στην ψηφιοποίηση και να αυξηθεί η παραγωγικότητα όπως πρέπει. γιατί τη ρομποτική και τα ρομπότ που έχουν και αυτά τη σπουδαιότητά τους μέσα στο πλαίσιο αυτής της έκθεσης πρέπει να στρέψουμε και σε αυτό το θέμα το βλέμμα μας και σε αυτό που αναφέρθηκε για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και τη διασυνδεσιμότητα. Αν δεν τα καταφέρουμε θα υπάρξουν πολλά προβλήματα στην ψηφιοποίηση και διαθροτικά προβλήματα και βλέπουμε ότι υπάρχει εδώ πολύ μεγάλη ανάγκη με ταχύτατους ρυθμούς να προχωρήσουμε για να ξεπεράσουμε τα προβλήματα και να υπάρξουν προ, προτάσεις για τη ρύθμιση που θα είναι σωστές για την ψηφιοποίηση και των επιχειρήσεων που με βάση τις υποδομές θα μπορέσουν έτσι να προχωρήσουν. Με αυτή την ευκαιρία θέλω να επισημάνω ότι είναι σημαντικό να επενδύσουμε στη διεύρυνση των υποδομών διότι χωρίς αποδοτική τέτοια υποδομή δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε την ε, ε, επίτευξη των στόχων για την ψηφιοποίηση. Για όλους αυτούς τους λόγους είναι σημαντικό η έκθεση να ασχοληθεί με τη θεματολογία των υποδομών, αλλά και με το νέο εργασιακό πλαίσιο, με την ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων συνολικά θα είναι αναγκαίο να αντιμετωπιστεί αυτό το νέο εργασιακό πλαίσιο. Χρειάζονται και μέτρα εκπαίδευσης, κατάρτισης από πλευράς παιδείας και στην τυποποίηση πρέπει να γίνουν πολλά και στην χρηματοδότηση και στην ενίσχυση. Ελπίζω ότι θα δώσει επαρκείς απαντήσεις σε όλα αυτά τα ερωτήματα η έκθεση. Ευχαριστώ. Πριν δώσουμε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δίνω το λόγο στην συνάδελφο Μαρτίνα Βέμπερ. Ευχαριστώ θερμά κυρία Πρόεδρε. Εδώ κάνουμε λόγο στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι η σπονδυλική στήλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σπονδυλική στήλη, 69% όλων των εργαζόμενων εργάζονται στις ΜΜΕ και πρόκειται στον πυρήνα για την διασυνδεσιμότητα, τη διασύνδεση όλων αυτών των επιχειρήσεων με τους μικρούς παρόχους τους και εδώ πρέπει να δούμε την παραγωγή και την δυνατότητα ψηφιοποίησης των μεθόδων παραγωγής. Υπάρχει όμως ο κίνδυνος εδώ να χάσουμε ένα βήμα. Η Τράπεζα Επενδύσεων ε, είδε πως ε, η κατάσταση πραγμάτων δίνει δυνατότητα να δούμε αν έχουν προετοιμαστεί επιχειρήσεις σωστά και βλέπουμε ότι σε σχέση με τη Γερμανία και άλλοι συνάδελφοι από άλλα κράτη-μέλη γνωρίζουν τα προβλήματα. Στη μελέτη αυτή οι πτυχές που αφορούν τη χρήση της ε, τεχνολογίας ε, και τις ψηφιοποίησεις ε, που δημιουργούν προβλήματα είναι πολλές σελίδες ε, ε, τα όσα απαριθμούνται. Δηλαδή, απουσία ενός ασφαλούς πλαισίου, μη επαρκής ταχύτητα, έλλειψη χρηματοοικονομικών δυνατοτήτων για επενδύσεις. Επιχειρήσεις λοιπόν για πολλούς λόγους βλέπουν ότι δεν μπορούν να, επιχειρήσουν, να επηρεάσουν τα πράγματα. Θέλουμε τη διασυνδεμότητα φυσικά να μην την επιβάλλουμε. Όμως παρακαλώ θα πρέπει σε ευρωπαϊκό επίπεδο να δημιουργήσουμε συνθήκες πλαίσιο που θα διευκολύνουν. Θα δώσουν δυνατότητα αυτές οι δυνατότητες μεταμόρφωσης ή στην πρακτική εφαρμογή να αποκτήσουν σάρκα και οστά. Και έτσι λοιπόν θα πρέπει να δούμε αυτά τα πράγματα στρεφόμενοι και προς την Επιτροπή. Διατυπώνουμε τώρα όλα αυτά σε σχέση με την αναθεώρηση για τα τηλεπικοινωνιακά και με την ε, ε, ιδιωτική και δημόσια πρωτοβουλία που θα πρέπει να συνδυάζεται και για τα ρομποτικά που θα έχουμε και την ψήφιση αύριο εδώ. Με αυτή τη σύντομη απαρίθμηση αναγνωρίζει κανείς ότι η ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων είναι ένα ιδιαίτερα οριζόντιο θέμα εγκάρσιο θέμα και γι' αυτό χαίρομαι για την περαιτέρω συζήτηση και συνεργασία μας. Ευχαριστώ Μαρτίνα. Έχουμε δύο παρεμβάσεις από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρώτη τη DG Connect. Ο κύριος Λέγκε έχει το λόγο. Έχετε το λόγο. Thank you, Chair. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Uh, Οι διάφορες παρεμβάσεις τόνισαν τη μεταμόρφωση που γίνεται στη βιομηχανία και την οικονομία αλλά και την κοινωνία. Όλα αυτά οι αλλαγές από την ψηφιακή τεχνολογία. Και είδαμε και ποια είναι η κλίμακα των προς αντιμετώπιση προβλημάτων. Το Κοινοβούλιο ανέλαβε αυτό το έργο και χαιρόμαστε. Το πακέτο που προτείναμε στις 19 Απριλίου, ενεστώτος έτους, για την ψηφιοποίηση, προσπαθεί να καλύψει τα περισσότερα σημεία, αν μην όλα. Δεν θα αναλύσω διεξοδικά τα προβλήματα που έχουν μπροστά μας, αλλά και τις τεράστιες ευκαιρίες που απορρέουν από την ψηφιακή μεταμόρφωση. Το πακέτο που προτείναμε εμπεριέχει πέντε βασικά τμήματα. Ξεκινάω από αυτό που αναφέρατε. Δεξιότητες, προσαρμογή του εργατικού δυναμικού, του εργασιακού περιβάλλοντος επίσης. Είναι σημαντικότατα αυτά. Αυτό σχετίζεται με τις διαφορές που αναφέρατε στην Ένωση. Τις διαφορές μεταξύ κρατών μελών, αλλά και μεταξύ περιοχών των κρατών. Σχετίζεται και με τις εταιρείε υψηλής τεχνολογίας που πηγαίνουν καλά και έχουμε αρκετές καλές στην Ευρώπη που πάνε καλά και τη διαφορά που έχουν με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις μεσαίες επιχειρήσεις που δεν είναι τεχνολογικά τόσο ανεπτυγμένες που θα πρέπει να προσαρμοστούν στις ψηφιακές αλλαγές και τις καινοτομίες. Οι δεξιότητες. Αυτό είναι κάτι που αφορά την εκπαίδευση, τη διαβίου μάθηση. Είναι κάτι που αφορά τα κράτη-μέλη. Υπάρχει περιθώριο, κατά την άποψή μας, συλλογικής προσπαθίας στην Ένωση για την προσαρμογή του εργασιακού περιβάλλοντος και του εργατικού δυναμικού στις αλλαγές, αλλά και του εκπαιδευτικού συστήματος μέσω της διαβίου εκμάθησης, να προσαρμοστούν όλοι οι τομείς στην ψηφιακή εποχή. Προτείναμε συνεργασία όλων των φορέων, κατών μελών, επαγγελματιών, εκπαιδευτών, επιχειρήσεων, συνδικάτων, να επανεξετάσουν το εκπαιδευτικό σύστημα και πώς εκπαιδεύεται ο κόσμος και το εργατικό δυναμικό. Δημιουργούμε μια συμμαχία η οποία επεκτείνεται μεταξύ των φορέων συμμαχία. Θέλουμε να επανεξετάσουμε όλες τις πτυχές που σχετίζονται με τις δεξιότητες και την προσαρμογή του εργατικού δυναμικού και θέλουμε να εφαρμόσουμε συγκεκριμένες δράσεις από αυτού για τις δεξιότητες. Στην ανακοίνωσή μας έχουμε συγκεκριμένες λεπτομέρειες δράσεις. Άλλη πτυχή, εμπιστοσύνη και το νομικό περιβάλλον που δημιουργεί την εμπιστοσύνη τονίζουμε δύο βασικά ζητήματα σημαντικότατα για τη βιομηχανία. Το θέμα των δεδομένων. Πώς χρησιμοποιούμε τα δεδομένα. Έχουμε ελεύθερη ροή δεδομένων και τη σχετική ανακοίνωση που προσπαθεί να τα καλύψει αυτά τα θέματα. Και θα επεξεργαστούμε και την χρήση των δεδομένων. Τι σημαίνει αυτό για τη βιομηχανία. Για ανώνυμα δεδομένα μιλάμε. Δεν μιλάμε για προσωπικά δεδομένα και την προστασία αυτών που καλύπτεται αλλού. Τι μπορεί να κάνει η βιομηχανία με τα δεδομένα, αυτό καλύπτουμε. Και η ασφάλεια των δεδομένων αυτών, που είναι σημαντικότατο. Και κάτι άλλο που σχετίζεται με την ε, εμπιστοσύνη είναι το θέμα των ευθυνών. Θέλουμε μεγαλύτερη αυτονομία, χρήση περισσότερων ρομπότ κλπ. Ε, προϊόντα, τεχνουργήματα κλπ. που παράγονται αυτόν τον τρόπο. Ρομπότ στο εργοστάσιο δημιουργούνται θέματα ευθυνών. Και η έκθεση του Κοινοβουλίου για τη ρομποτική είναι διεξοδική για αυτά τα ζητήματα. Δύο-τρία βασικά στοιχεία της ρυθμιστικής προσαρμογής που προτείνουμε είναι αυτά. Είναι σημαντικότατα. Τα αναφέρατε κι εσείς άλλωστε. Και στις παρεμβάσεις και στην έκθεση. Και κάτι άλλο εξίσου σημαντικό. Καινοτομία. Θέλουμε καινοτομία να φτάνει σε όλες τις βιομηχανίες, ανεξαρτήτως μεγέθους και τόπου εγκατάστασης. Πρωταρχικός στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι αυτός. Οποιαδήποτε βιομηχανία ή οσδήποτε τομέας, εταιρεία ή οδήποτε είδους και μεγέθους να αφελείται και να δημιουργεί καινοτόμα προϊόντα με υψηλή προστιθέμενη ε, αξία χρησιμοποιώντας σωστά τους διαθέμενους πόρους και να υπάρχει σωστή προσαρμογή στις αλλαγές. Αυτό το κομμάτι περί καινοτομίας. Εμπεριέχει δύο στοιχεία. Πρώτον, η τεχνολογία πρέπει να είναι διαθέσιμη οπουδήποτε. Να μπορεί να τις χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις. Και προτείνουμε κύμα επενδύσεων και κέντρα γνώσεων και δεξιοτήτων. Εκεί πρέπει να κινηθούν τα κράτη-μέλη και οι περιφέρειες. Και από πλευρά Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής θα διαθέσουμε χρήματα από τους στόχους 2020 που θα εξασφαλίζει διασυνδεσιμότητα των κέντρων αυτών. Θέλουμε να στηρίξουμε και τον πειραματισμό σε διασυνοριακό επίπεδο. Τι μας λένε οι επιχειρήσεις γιατί διστα... και γιατί διστάζουν τα νέα μετά, ότι θέλουν να κάνουν δοκιμή, θέλουν να κάνουν πειράματα πριν πραγματικά ε, ενστερνιστούν κάτι καινούριο. Αυτό θέλουμε να κάνουμε, να αυξήσουμε τον πειραματισμό που είναι διαθέσιμο σε όλες τις επιχειρήσεις. Ούτως ώστε να δοκιμάσουν και να προωθήσουν την ψηφιακή καινοτομία. Αυτά περί καινοτομίας. Δεύτερον, πώς μπορούμε να ηγηθούμε στο ψηφιακό τομέα στην Ευρώπη. Έτσι η βιομηχανία μας θα μπορεί να παράξει προϊόντα με μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι έχουμε στοχευμένη προσπάθεια, έρευνα ανάπτυξη, πειραματισμό σε μεγάλη κλίμακα, τυποποίηση. Πολύ σημαντικό αυτό. Και μετά πλήρης χρήση και παραγωγής τεχνολογίας σε βασικούς τομείς οικονομίας επιτάχυνση της αναπτύξεως στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, αυτόματη οδήγηση κλπ, τηλεπικοινωνία, 5G, ε, υπολογιστική τεχνολογία, ε, πώς μπορούμε να παράξουμε προϊόντα όσον αφορά την πληροφορική πιο σύγχρονα και πιο παραγωγικά, πρέπει να ηγηθούμε στην Ευρώπη. Πρέπει να γίνουν προσπάθειες γι' αυτό σε όλα τα επίπεδα. Πέμπτο, σημαντικότατο. Αυτό που αναφέρατε κι εσείς, παραδοσιακή βιομηχανία. Όλα τα κράτη-μέλη να εφαρμόζουν τις πρωτοβουλίες τους. Έχουμε 11 κράτη-μέλη που κάνουν πρωτοβουλίες στον τομέα αυτό. Θέλουμε η ψηφιοποίηση της βιομηχανίας να λάβει η χώρα μέσω πρωτοβουλίων σε όλα τα κράτη-μέλη. Και έχουμε δημιουργήσει κατάλληλο πλαίσιο συντονισμού Αυτά προτείναμε, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, όλα αυτά μαζί με τέξη του Κοινοβουλίου ελπίζουμε ότι θα μας οδηγήσουν να ακινηθούμε σε κατεύθυνση. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα εδώ να διευκρινίσω. Σας ευχαριστώ που πήρατε το λόγο από την αρμόδια Γενική Διεύθυνση της Επιτροπής. Κοιτάξτε, έχουμε ξεπεράσει το χρόνο μας. Θα δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο τώρα της Γενικής Διεύθυνσης για την Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Uh, Από πλευρά τη βιομηχανία θα πρέπει να πω ότι η Ευρώπη έχει μια ηγετική θέση σε πολλού τομεί όπω την αυτοκίνητοβιομηχανία και την ιατρική τεχνολογία. Για να διατηρήσουμε όμω αυτή την ηγετική θέση πρέπει να εξυγχρονίσουμε τις παραγωγικές μας δραστηριότητες και γι' αυτό το πακέτο αυτό θα βοηθήσει πολύ την ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης. Νομίζω ότι η προστιθέμενη αξία των πραγματικών ψηφιακών τεχνολογιών είναι η σύγκλησή τους με τις υπόλοιπες τεχνολογίες και τα κοινοτέωμα μοντέλα πρότυπα παραγωγής. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα τονώσει την διεθνή ανταγωνιστικότητά μας. Αυτή η ψηφιακή αλλαγή θα έλεγα επηρεάζει όπως είπατε όλες τις βιομηχανίες, ε, τις τράπεζες, ε, την αυτοκινητοβιομηχανία και απαιτείται καλύτερη συνεργασία ανάμεσα στους κατασκευαστές από τη μία των διαφόρων τομέων και την ψηφιακή βιομηχανία. Τώρα για την ανακοίνωση σχετικά με τα κοινά μέτρα και σταθμά και είναι κάτι στο οποίο αναφερθήκατε αρκετοί από εσά. Πολλοί τομεί τη οικονομία εξαρτώνται από τι ψηφιακέ ε, αυτές τεχνολογίες που αλλάζουν με μεγάλη ταχύτητα. Τα σύνορα ανάμεσα στην παραδοσιακή ε, πληροφορική δραστηριότητα και ε, την τεχνολογία, τα σύνορα μερικές φορές είναι θολά. Απαιτείται λοιπόν διαλειτουργικότητα έτσι ώστε οι ψηφιακές τεχνολογίες να μπορούν να λειτουργήσουν και στο μέλλον. Η ανακοίνωση αποτελείται από δύο πυλώνες. Πρώτον, ε, η ιεράρχηση πέντε πυλώνων που θεωρούνται κατεπήγοντος ε, ε, όπως το cloud computing, η συλλογή δεδομένων, η συντήρηση συστημάτων και άλλοι τομείς στους οποίους απαιτείται δράση άμεσα. Η δράση σε αυτούς τους τομείς θα επιταχύνει την ψηφιοποίηση και θα επηρεάσει την ανταγωνιστικότητα στην ηλεκτρονική υγεία, τα FEE e συστήματα μεταφορών, τα αυτόματα αυτοκινούμενα οχήματα και την κατασκευή μηχανών βιομηχανίας, για τη βιομηχανία. Έτσι θα μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε, να, να εκρίνουμε τους τύπους των μηχανών που χρησιμοποιούνται και χρησιμοποιώντας το ευρωπαϊκό σύστημα κοινών μέτρων ε, θα έλεγα θα μπορέσουμε να συνεισφέρουμε στη διαλειτουργικότητα αυτή. Θα σας ενημερώσουμε για την πρόοδο, θα ενημερώσουμε επίσης και τους εκπροσώπους των βιομηχανικών και τις οργανώσεις ε, των κοινών προτύπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα δώσω το λόγο σύντομα τώρα στον κύριο Μπιούτι Κόφερ, ο οποίος ε, βιάζεται γιατί πρέπει να ταξιδέψει. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τις ακριβείς ε, εξειδικευμένες προτάσεις τους. Προσβλέπω στη συνεργασία μεταξύ μας και ευχαριστώ την Επιτροπή γιατί επανέλαβε αυτά τα οποία γνωρίζαμε. Ε, Σας ευχαριστώ όλους. Αφήνω την Προεδρία στον Πρόεδρό μας, τον κύριο Μπούσεκ και πιστεύω θα κάνει έξοχη δουλειά. Niente, figurati, it's a pleasure. Good morning, ladies and gentlemen. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Καλημέρα συνάδελφοι. We've got next. Πάμε στο επόμενο σημείο της ημερησίας διατάξεως των παριθμών 5 καινοτόμα φάρμακα και σχετική πρωτοβουλία, κοινή σύμπραξη στα πλαίσια του ορίζοντα 2020 και της υλοποίηση αυτού του στόχου. Παρουσίαση από τον εκτελεστικό διευθυντή της IMI, τον κύριο Πιέρ Μελιά. Επιτρέψτε μου να πω μερικά λόγια στην αρχή. Σαν αρμόδια επιτροπή Έχουμε καθήκον συνεχώς να αξιολογούμε την υλοποίηση των προγραμμάτων. Αν έχουν εμφανιστεί νέα προβλήματα, εάν χρειάζονται νομοθετικές ή δημοσιονομικές αλλαγές. Σε αυτό το πλαίσιο ε, είναι πολύ σημαντική η παρουσίαση. Η IMI είναι μία από πολλούς ε, μία από τις πολλές συμπράξεις ιδιωτικού και δημόσιου τομέα που εφαρμόζουν τα πλαίσια ε, του ε, Ίζοντα 2020 σύμφωνα με το άρθρο 187. Η IMI δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 μετά από επιτυχείς διαπραγματεύσεις στο Ευρωκοινοβούλιο στο τέλος της προηγούμενης θητείας στα πλαίσια ενός πακέτου ε, διαφόρων συμπράξεων του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα. Θα παρακαλούσα λοιπόν τον κύριο Γενικό Διευθυντή να παρουσιάσει ίσως σύντομα το θέμα αυτό. Είναι η μεγαλύτερη σύμπραξη στον κόσμο ιδιωτικού δημοσίου τομέα όσον αφορά αυτό το, το, το τομέα των επιστημών. να μας πει κάποια πράγματα. Λοιπόν, έχετε το λόγο να μας παρουσιάσετε το όλο θέμα. Ευχαριστώ κύριε Μπούζεκ, μέλη του Ευρωκοινοβουλίου. Ευχαριστώ πολύ που με επιτρέπετε να σε ενημερώσω σχετικά με την πρωτοβουλία για τα καινοτόμα φάρμακα. Το Ευρωκοινοβούλιο ήταν πολύ σημαντικό για να δημιουργηθεί αυτή η συνεργασία, αυτή η σύμπραξη και χαίρομαι που έρχομαι εδώ να σας ενημερώσω. επενθυμίσω κάτι εν συντομία. Πρόκειται περί πολύ μεγάλης πρωτοβουλίας με ένα προϋπολογισμό 5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Είναι σύμπραξη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας της Φαρμακοβιομηχανίας και διαφόρων ε, συνδέσμων του τομέα η φαρμακοβιομηχανία συμβάλλει εις είδος και δεν λαμβάνει χρήματα της ε, Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Τα χρήματα πηγαίνουν στο, στους τέρους μας του δημοσίου στη σύμπραξη αυτή. Γιατί χρειαζόμαστε την IMI στο χώρο των καινοτόμων φαρμάκων. Η έρευνα και η ανάπτυξη είναι περιπλοκότατη, ελοχεύουν πολύ κίνδυνοι, μακροχρόνια, δαπανηροί. Οι βιολογικοί μηχανισμοί ε, των ασθενειών ε, είναι πολύ περίπλοκη, αλλά και η επιστημονική πρόοδος είναι πάρα πολύ σημαντική, εντυπωσιακή και έχει μεγάλο αντίκτυπο όχι στον αφορά την κατανόηση των ασθενειών, αλλά και στο σχεδιασμό των κλινικών δοκιμασιών και να διευκολύνουμε και την πρόσβαση των ασθενών στην καινοτομία. Εγκαίρως. Έξοχη η έρευνα σε όλο τον κόσμο για πολλές ασθένειες. Παρ' αυτά δεν έχουμε αρκετά νέα αντιβιωτικά για την αντιμετώπιση ε, της αντιστάσεως των μικροβίων στα αντιβιωτικά. Δεν έχουμε θεραπεία για το διαβήτη, ε, για την άνοια. Λοιπόν, ε, υποστηρίζουμε ανάπτυξη προϊόντων σε ένα ευρύ φάσμα και την καινοτομία. Εντοπίζουμε μεθόδους διαγνωστικής, φάρμακα, δοκιμές, εξετάζουμε τα θέματα ασφαλείας των καινοτόμων προϊόντων και ελπίζουμε ότι γίνεται δέωσα προσαρμογή των διαδικασιών για την αύξηση αποδοτικότητας. Στη χρηματοδότηση τώρα των προγραμμάτων ε, δημιουργούμε ένα νέο οικοσύστημα, νέο είδους οικοσύστημα ε, ιδιωτικής και δημόσιας σφαίρας. 9.000 ε, ερευνητές, πάνω από 9.000 ερευνητές ε, συμμετέχουν, πάρα πολλές ομάδες, πάνω από 202 από 200 μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ομάδες ασθενών που είναι πολύ σημαντικοί. 970 ομάδες πανεπιστημιακών και δημιουργούμε αυτό το οικοσύστημα στην Ευρώπη στην IMI έχουμε διανύμει την χρηματοδότηση όπως βλέπετε. Βλέπετε στο γράφημα πώς διανέμονται τα πόροι του IMI-1 και οι αρχές του IMI-2. Βλέπετε τις διάφορες ασθένειες. Βλέπετε ένα μεγάλο κομμάτι στις μεταδοτικές ασθένειες μέσω πολύ μεγάλου προγράμματος που εφαρμόζουμε για την καταπολέμηση της αντιστάσεως των μικροβίων στα αντιβιωτικά, που είναι απειλή. Ένα-δύο λεπτά προς το τέλος θα σας δώσω κάποια παραδείγματα της δουλειάς που κάνουμε. Πρώτα απ' όλα βλέπετε όσον αφορά την αντίσταση των μικροβίων στα αντιβιωτικά ε, που είναι μια αυξανόμενη απειλή, θα διαβάσετε τη σχετική έκθεση και προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα σε πολλά επίπεδα ερευνών. Πρώτο επίπεδο, πώς τα νέα φάρμακα τα βάζουμε στα βακτήρια που θέλουμε να είναι στόχοι μας Δεύτερον, πώς μπορούμε να δώσουμε τη δυνατότητα, να αυξήσουμε την αποδοτικότητα του να διατίθενται νέα φάρμακα στις κλινικές δοκιμές. Συμμετέχουν πολλές μικρόμεσες επιχειρήσεις. Η διαδικασία των κλινικών δοκιμών είναι χρονοβόρα, χρειάζεται εξειδικευμένα δίκτυα, τα οποία τα δημιουργούμε σε όλη την Ευρώπη. Και τέλος, επίσης προσπαθούμε να δημιουργήσουμε νέα επιχειρηματικά μοντέλα, ούτως ώστε να δώσουμε κίνητρα στη βιομηχανία να επενδύσει σε αυτό το τομέα που βέβαια ε, είναι ένας τομέας με πάρα πολλά προβλήματα και προκλήσεις. Μετά η ασθένεια Alzheimer και η άνοια, δεν χρειάζεται να περιγράψω το θέμα εδώ. 50 εκατομμύριο άνθρωποι ε, ασθενούν από αυτά και με τη γύρανση του πληθυσμού που αυξάνεται το ποσοστό των ηλικιωμένων στην κοινωνία μας, αυξάνονται και τα προβλήματα. Εδώ βλέπετε, δεν προσπαθούμε να βρούμε μόνο τα αίτια της άνοιας, αλλά και ποιοι είναι οι κίνδυνοι που σχετίζονται με την άνοια, δηλαδή ποιοι έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να πάθουν άνοια, πώς μπορούμε εγκαίρως να παρέμβουμε πριν ε, εγκατασταθεί ε, αμετάκλητα η ασθένεια και πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ε, και άλλες τεχνολογίες, όχι μόνο την ιατρική, αλλά τεχνολογία απεικόνησης κλπ. Στις 8 Νοεμβρίου, ο κύριος Μαραγκάλ και συνάδελφοι θα φιλοξενήσουν μια εκδήλωση όσον αφορά τα προγράμματα της AMI για το Alzheimer και καλέσαμε και το πρόγραμμα για τον ανθρώπινο εγκέφαλο που χρηματοδοτείται τα DG Connect, άρα βλέπετε ότι είναι εγκάρσια, οριζόντια προσέγγιση όσον αφορά το ψηφιακό θέμα που συζητήσατε σχετικά με τις πιο πρόσφατες έρευνες για το Alzheimer. Μετά κάποια εγκάσια θέματα, οριζόντια θέματα, όπως η ασφάλεια των φαρμάκων, είναι αρκετά σημαντικό το θέμα, η αντιδράση παρενέργειες των φαρμάκων, οι παρενέργειες δημιουργούν θνησιμότητα, προβλήματα κινητικότητας κλπ. και θα πρέπει έγκαιρα να δούμε πώς μπορούμε να προβλέψουμε ε, την τοξικότητα των μορίων πριν αυτά ε, μπουν στον οργανισμό των ανθρώπων. Έχουμε δύο προγράμματα, έχουμε το e-tox, το οποίο ουσιαστικά οδηγεί σε μεγαλύτερη συνεργασία της φαρμακοβιομηχανίας. Συλλογικά παράγουν δεδομένα σε ομάδες δεδομένων. Εδώ είναι ένα από τα μεγάλα προγράμματα περί συλλογής δεδομένων δεν θα μπορούσαμε χωρίς το IMI να τα πετύχουμε αυτά, διότι όλοι ε, αθρίζονται τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα. Μπορεί κανείς λοιπόν να δοκιμάσει το νέο φάρμακο μέσω της βάσης δεδομένων, βάση κριτηρίων να ελέγξει το νέο φάρμακο όσον αφορά την τοξικότητα του φαρμάκου και αυτό συμβάλλει κατά πολύ στην μείωση της χρήσης ζώων στην έρευνα. Τελικά, Έχουμε ε, πολύ μεγάλα προγράμματα σε αρχικό στάδιο αναπτύξεως φαρμάκων. Εδώ αφορά την χρήση μεγάλη συλλογή συστατικών. Πριν αυτή η συλλογή θα ήταν πάρα θα καλύπτεται από μυστικότητα. Σήμερα 7 εταιρείε ομαδοποιούν αυτά τα στοιχεία τα στατικά, ενημερώνουν τους πανεπιστημιακούς, ε, και δημιουργούν μια ε, τεκμηρίωση που είναι πάρα πολύ ποιοτική, πολύ ογκώδης και πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν και να ενημερωθούν. Και είναι η μεγάλη επιτυχία του European Lead Factory που δημιουργήσαμε με, και εκπονούμε και πολλά εμπορικά, εμπορικές, ε, επιστημονικές μελέτες, άρθρα κλπ. Ε, όχι μόνο δημιουργούμε αριστεία στον τομέα της έρευνας, αλλά επηρεάζουμε και το ρυθμιστικό κομμάτι της εξίσωσης και το επιχειρηματικό. Πολλά από τα προγράμματά μας αφορούν τις αγορές, βιολογικές αγορές, και τους βιολογικούς δείκτες που είναι απαραίτητοι για τη λειτουργία των υπηρεσιών ελέγχου φαρμακευτικών ουσιών. Εμείς προσπαθούμε εξ αρχής να παρακολουθήσουμε τις διαδικασίες αυτούς και να εμπλέξουμε όχι μόνο τους ασθενείς και όχι μόνο τις ρυθμιστικές αρχές, αλλά και εκπροσώπους του ιατρικού κόσμου και άλλα σώματα που μας διευκολύνουν να ευθυγραμμίσουμε τις διαδικασίες αυτές. Το θέμα είναι πώς θα μπορέσουμε να στηρίξουμε στην παρούσα φάση τα σύνολα δεδομένων τα οποία έχουν συλλεχθεί στο παρελθόν, τα ιδρύματα τα οποία έχουν επίσης δημιουργηθεί με βάση τα δεδομένα αυτά και χρηματοδοτούνται από τον φαρμακευτικό και άλλους τομείς. Γιατί προβλέπεται ότι θα έχουν τεράστια προστιθέμενη αξία στην προσπάθεια η οποία γίνεται. Και τέλος, και θα προσπαθήσω να κλείσω, ε, έχουμε, εντοπίσει την προσοχή μας στις ομάδες των ασθενών. Είναι τμήμα ε, των ε, σχεδίων μας, των προγραμμάτων μας. Το JDRF είναι εταίρος στην προσπάθεια για το διαβήτη. Έχουμε επίσης αντίστοιχες προσπάθειες και για την άνοια κτλ. κτλ. Έχω λίγο, δεν έχω μάλλον χρόνο στις ιστοσελίδες μας. Έχουμε πάρα πολλές πληροφορίες για όλους. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Very, very much. Τον κύριο Μελιέ. Η κυρία Γκροστέτ θέλει να θέσει κάποιες ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ, λέει η κυρία Γκροστέτ. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον Γενικό Διευθύντη της IMI, να τον συγχαρώ για την εξαιρετική δουλειά την οποία έχει κάνει από το 2015. Η παρέμβασή σας ήταν μεν συνοπτική, αλλά δείχνει το ενδιαφέρον που έχει ε, το IMI. Δεν είναι εύκολο να πείσει κανείς. Εγώ ήμουν εισηγήτρια για την δημιουργία του IMI και μετά τα εισηγήτρια για το IMI2. Και γνωρίζω ποιες είναι οι κριτικές οι οποίες ασκούνται και είναι αφεμελίωτες κατ' με... απέναντι σε αυτή την μορφή συνεργασίας του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Πάρα πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι φοβούνται αυτού του είδους τις εταιρικέ σχέσεις. Εγώ αντίθετα πιστεύω ότι πρόκειται για μια ουσιαστική πρωτοβουλία Πρόκειται για ένα ισχυρότατο μήνυμα το οποίο δίδει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα της ιατρικής καινοτομίας. Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο άλλωστε μας απασχόλησε και στην Επιτροπή Ένβη σήμερα το πρωί, η πρόσβαση στα φάρμακα και στην καινοτομία των ασθενών. Ακούγοντας και τους περισσότερους από τους συναδέλφους, ε, βλέπω ότι απαιτείται παιδαγωγική μάλλον δραστηριότητα έτσι ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε ακόμα περισσότερο την ιατρική καινοτομία. Συγχαρητήρια λοιπόν για τις ε, ενέργειες του IMI, χάρη στον ορίζοντα 2020 και την πρωτοβουλία για τα καινοτόμα φάρμακα, η Ευρώπη αποστέλει ένα ξεκάθαρο και ισχυρότατο μήνυμα. Δεν γίνεται συχνά κάτι τέτοιο σχετικά με αυτά τα οποία κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να πούμε λοιπόν ότι σήμερα μπορούμε να κινητοποιήσουμε τα απαιτούμενα οικονομικά μέσα έτσι ώστε να δημιουργήσουμε τις συνέργειες τις απαραίτητες για την καινοτομία. Υπάρχουν δύο ερευνητικοί τομείς στους οποίους αναφερθήκατε και είναι τμήματα των προτεραιοτήτων του IMI2. Πρώτον, Alzheimer, άνοια όπως το είπατε, και ό,τι έχει σχέση με τις ασθένειες αυτού του τύπου και επίσης από την άλλη αντίσταση στα α, αντιβιωτικά και τα αντιμικροβιακά φάρμακα. Έχω μία ερώτηση πάνω σε αυτά τα δύο φάρμακα, Αλτσχάιμερ από τη μία και αντίσταση στα αντιμικροβιακά. Μπορείτε να μας δώσετε κάποια περισσότερα στοιχεία για τα αποτελέσματα στα οποία καταλήγετε γιατί όλοι ενδιαφέρονται γι' αυτό. Ευχαριστώ κύριε Αγκρός Τέτ. Ο κύριος Πόχε καλή σας μέρα, πρόεδρε, κύριε Διευθυντά, συνάδελφοι. Διευθυντά, θέλω να σας ευχαριστήσω. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας. Ενδιαφέρομαι πάρα πολύ στην πρωτοβουλία IMI EMI, καθώς επίσης και όσον αφορά και την Επιτροπή Ελέγχου. Δηλαδή, για όλες τις κοινέ τέτοιες επιχειρήσεις, ε, πρωτοβουλίες και χαίρομαι και για τα αποτελέσματα ε, αυτών των πρωτοβουλίων τους τελευταίους μήνες και μάλιστα με έναν ε, τρόπο που είχε προβλέψει και προωθήσει θέματα για τον ορίζοντα 2020 για παράδειγμα και κοινέ τέτοιες πρωτοβουλίες που πρέπει να λυθούν υπόψη για παράδειγμα, σε σχέση με το ποσοστό σφάλματος ε, όσον αφορά την διαχείριση κοινών τέτοιων πρωτοβουλειών και προγραμμάτων. Κοινωνικονομικές επιπτώσεις. Μια άλλη ανάλυση που πρόσφατα λάβαμε. Δύο ερωτήσεις θα ήθελα να διατυπώσω. Ποια είναι η μεγαλύτερη, η μέγιστη πρόσθετη αξία για προγράμματα τα οποία δεν στοχεύουν σε κλινικές ή βασικές έρευνες για παράδειγμα εκπαίδευση, κατάρτιση σε σχέση με την ε, ε, ε, δημιουργία νέων φαρμάκων, φάρμα και την έρευνα γενικότερα. Τα τελευταία δύο χρόνια οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είχαν συμπεριληφθεί περισσότερο, 16% ήταν για παράδειγμα νομίζω το 2015 και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την ε, συμμετοχή και ε, εμπλοκή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε τέτοιου είδους ε, δράσεις. Δυστυχώς όμως δεν υπήρξε μια τέτοια σημαντική αύξηση. Τι θα θεωρούσατε το μεγαλύτερο πρόσκομα για τη συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Thank you. And, uh, firstly, Ευχαριστώ. Καταρχάς, βάσει των σχολείων που ακούστηκαν από κάποια πράγματα περί επιτευμάτων του IMI μέχρι τώρα και των προσδοκιών για άλλα επιτεύγματα. Όλοι έχουμε ευθύνη να κοινοποιούμε στους πολίτες καλύτερα τα όσα συμβαίνουν. Είτε είναι για το Alzheimer, για το διαβήτη, για άλλη ασθένεια. να δείξουμε ότι ωφελούνται οι ασθενείς από τη δουλειά που κάνετε. Και το άλλο για τι συμπράξεις ιδιωτικού δημόσιου τομέα σε αυτό το τομέα είναι ένα καλό παράδειγμα. Επιλύει τα προβλήματα τα παλιά της αγοράς και δίνει αποδεδειγμένα προστιθέμενη αξία στον τομέα των φαρμάκων. Ερώτηση. Πώς να το πω τώρα. Γνωρίζω ότι υπάρχουν πανεπιστήμια στην περιοχή μου, στον Ηνωμένο Βασίλειο, που ε, συμμετέχουν ενεργά στις προσπάθειες του IMI. Ιατρική έρευνα, φιλανθρωπικούς οργανισμούς κλπ. Ε, ξέρω ότι όλοι αυτοί εκτιμούν τα μάλα αυτές τις προσπάθειες και συμμετέχουν. Πώς βλέπετε εσείς το ρόλο της έρευνας ε, και των επιστημών στην Ηνωμένο Βασίλειο. Πώς συμβάλλουμε στις προσπάθειες ε, του IMI σαν Ηνωμένο Βασίλειο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ζωρίνιο έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και να συγχαρώ ε, τον παρουσιαστή για την έκθεση που παρουσίασε. Να συγχαρώ για το έργο της η πρόσβαση στα καινοτόμα φάρμακα έχει θεμελιώδη σημασία. Σε σχέση με, τις προόδους, με την πρόοδο πρέπει να εξευρεθούν και νέες απαντήσεις και νέες δυνατότητες. Θα πρέπει επίσης να ευρεθούν, εξευρεθούν απαντήσεις ε, σε σχέση με τις προηγούμενες ε, ε, απαντήσεις, την μη ύπαρξή τους. Ε, ο συνδυασμός ε, των ε, δυνατοτήτων αυτών ιδιωτικών και δημόσιων είναι πολύ σημαντικό για να καταλήξουν τα ευρωπαϊκά κονδύλια στους πολίτες για να ζήσουν και να βιώσουν ότι εποφελούνται άμεσα από αυτά τα κονδύλια. Ωστόσο αυτό θέλω να θέσω μια ερώτηση αντίστροφη κάπως. Όταν συζητείτε αυτή η θεματολογία στη χώρα μου, για παράδειγμα, με τα καινοτόμα φάρμακα, πάντα τίθεται το ερώτημα της επίπτωσης στις τιμές. Ποια επίπτωση θα έχουν οι τιμές. Με άλλα λόγια δηλαδή, αφενός, μέχρι ποιο σημείο αυτά τα καινοτόμα φάρμακα μπορεί να οδηγήσουν στο να λόγω του κόστους να καταρρεύσουν τα ε, συστήματα περίθαλψης ε, και άλλου είδους φάρμακα να είναι διαθέσιμα ή αν δεν υπησέλθουν στο σύστημα αυτό πολλά άτομα θα μείνουν εκτός της δυνατότητας να χρησιμοποιήσουν αυτά τα φάρμακα. Διαρωτώ με πώς αυτό όλο το συνολικό σύστημα θα είχε επιπτώσει στη διαμόρφωση των τελικών τιμών των φαρμάκων. Ευχαριστώ. κύριος Κόχλιτσεκ παρακαλώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε έχω κάποιες ίσονος σημασίας ίσως ερωτήσεις. Αναφέρθηκαν οι εξαιρετικές επιτυχίες που σημειώθηκαν. Πολλοί ερωτούν και ποια είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τι καταφέρνει. Ιδού λοιπόν το πεδίο και η απάντηση. Ερώτησή μου πέρα από την νόσο Αλτσχάιμερ και τον ιδιαίτερα περίπλοκο χαρακτήρα της διότι και εγώ ο ίδιος ε, έχω ε, συμμετάσχει σε αυτή την προσπάθεια και γνωρίζω ότι πόρο απέχουμε από την ε, τελική λύση. Επίσης για άλλες ασθένειες υπάρχει μεγάλη πορεία να καλυφθεί. Ερώτηση, θα εμπλακείτε στα ρομποτικά Πολλοί έχασαν τη θέση απασχόλησής τους από τους εργαζόμενους λόγω της ρομποτικής και είναι ένας τομέας που έχει πολύ μεγάλη εμβέλεια. Κα, καρκίνος, άλλο πεδίο. Υπάρχει για παράδειγμα και ο καρκίνος της μήτρας που ε, γίνονται πολλές έρευνες και υπάρχουν και πολλοί άγνωστοι συντελεστές και στοιχεία και άλλοι τομείς ε, που ε, μπορεί να σκεφτεί κανείς ε, ορθοπαιδική για παράδειγμα για την, ε, τα προβλήματα των ισχύων και την αντικατάσταση με συγκεκριμένο τρόπο αυτών των αρθρώσεων. Ευχαριστώ. Well, thank you very much. And it's, uh, uh, very all uh, excellent questions that are... Έξοχες ερωτήσεις. Θα απαντήσω μία-μία. Ευχαριστώ κυρία Γκροστέτ για την παρέμβασή σας. νομίζω ότι αυτό που μπορέσαμε να κάνουμε είναι να καλέσουμε μικρές επιχειρήσεις, μικρομεσαίες επιχειρήσεις να έρθουν στο τραπέζι ενός πολύ εμπειρού πάνελ για να τους δοθούν συμβουλές για το αν πρέπει να προωθήσουν κάποια μόρια ή όχι. Έχουν μεγάλη εμπειρία αυτοί στην ΕΜΑΡ και μπορούν πολύ εύκολα να κατευθύνουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο για την AMR υπάρχει όχι μόνο ένα ευρωπαϊκό δίκτυο αλλά και παγκόσμιο δίκτυο και ήταν ένα από τα προγράμματα που αποκτά διεθνή απόχρωση λόγω των τεκτονωμένων στις ΙΠΑ και αλλού. Πρέπει να ενώσουμε τις κουκίδες σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι εικόνα. Δεν είναι μόνο ευρωπαϊκό το πρόβλημα, αλλά παγκόσμιο. Για την όσο άλτσχαϊμερ δύο πράγματα. Προσπαθούμε να αποκρυπτογραφήσουμε διάφορα είδη Αλτσχάιμερ διότι Alzheimer δεν είναι μία ασθένεια. Έχει, περιέχει πολλούς τύπους. Οπότε θα δημιουργήσουμε υποκατηγορίες. Και είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι θα βγει. Διότι αυτή η διαστρωμάτωση των ε, εκφάνσεων της ασθένειας θα μας οδηγήσει σημαντικά συμπεράσματα. Και έχουμε ασθενείς τους οποίους θα μπορούμε να πλησιάσουμε πριν εγκατασταθεί μόνιμα η ασθένεια το ΣΥΠΗΝ και να μπορούμε να κάνουμε κάτι για αυτούς και να επιτεθεί πρόοδος. Κοινωνικο-οικονομικός αντίκτυπος, κύριε Πόχε. Εκπαίδευση, το θέμα της κατάρτισης και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έχετε δίκιο λοιπόν ότι το θέμα της κατάρτισης εδώ και η συμπερίληψή του στο χώρο της επεξεργασίας και της έρευνας για τα καινοτόμα φάρμακα είναι πολύ σημαντικό. Το θέμα δεν είναι μόνο να εκπαιδεύσουμε τον χώρο αυτό, για τον χώρο αυτό τους ειδικού επί της υγείας, αλλά και τους ασθενείς, γιατί οι φωνές των ασθενών έχουν αρχίσει και ακούγονται όλο και περισσότερο και ένα από τα προγράμματά μας είναι κάποια πρότυπα σεμινάρια εκπαίδευσης ασθενών. η εμπλοκή των μικρομεσαίων στα πλαίσια του IMI1 ήταν γύρω στο 60%. Τώρα είμαστε χαμηλότερα. Ενδιαφερόμαστε λοιπόν στο να δούμε ποια είναι τα προβλήματα τα οποία εμποδίζουν την συμμετοχή των μικρομεσαίων να εμπλακούν περισσότερο, να κατανοήσουν τα πλαίσια για την πνευματική ε, ιδιοκτησία δεν είναι τόσο περίπλοκα τα θέματα, νομίζω ότι αδίκως φοβούνται πολύ. Πολλές μικρομεσαίες ε, διστάζουν να εμπλακούν σε συνεργασία με μεγάλα κονσόρτια βιομηχανικά στον τομέα της φαρμακευτικής. Για την κυρία Μούντι, η ερώτησή σας είναι πολύ σημαντική για μας. Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι η πρώτη χώρα που ωφελείται από το IMI. Εκτιμούμε ιδιαίτερα επίσης αυτό το οποίο κάνουν οι επιχειρήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα πανεπιστήμια και οι ομάδες των ασθενών. Είναι πάρα πολύ παραγωγικές, όριμες και εμπλέκονται συνεχώς. Το Ηνωμένο Βασίλειο λοιπόν είναι σημαντικότατο για μας και ελπίζω να βρούμε έναν τρόπο να συνεχίσουμε την συνεργασία. Προς το παρόν εμείς εφαρμόζουμε την αρχή business as usual. Συνεχίζεται η προσπάθεια έτσι όπως τη γνωρίζαμε μέχρι τώρα, αλλά πάντως σας ευχαριστούμε για τα ερωτήματά σας. Από τον κύριο Ζωρίνιο για την τιμολόγηση. Αυτό είναι ένα πολύ περίπλοκο θέμα, ένα θέμα στο οποίο δημιουργούνται δυσκολίες. Ξέρετε ότι η τιμολόγηση των φαρμάκων δεν είναι ευρωπαϊκή αρμοδιότητα. Είναι κάτι το οποίο ανήκει στα κράτη-μέλη μεμονωμένα και εκεί συμβαίνουν οι διαπραγματεύσεις. Νομίζω ότι αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε στα πλαίσια του IMI είναι να καταστήσουμε τη διαδικασία αυτή για την έρευνα και την καινοτομία να γίνει πιο αποτελεσματική και ελπίζουμε ότι αυτό θα οδηγήσει σε ευθυνότερα φάρμακα. Το σύνολο της ιδέας, αν θέλετε, της τροματοποίησης που οδηγεί στο προσωπικό φάρμακο, αυτό μπορεί να βοηθήσει να υπάρξουν πιο στοχευμένες θεραπείες αλλά μια τέτοια διαδικασία δεν θα λειτουργήσει αν τα συστήματα υγείας δεν μπορούν να πληρώσουν για αυτά τα φάρμακα. Η προσπάθειά μας λοιπόν είναι τέτοιου τύπου έτσι ώστε να αυξήσουμε εξ αρχής την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας και να μειώσουμε το κόστος. Σήμερα δυστυχώς οικονομικά δεν είναι κάτι το ιδιαίτερα παραγωγικό. Και τέλος υπήρξαν και αρκετές ερωτήσεις για άλλα θέματα. Έχουμε και στον τομέα του καρκίνου κάνει αρκετές προσπάθειες, θα εμπλακούμε ακόμα περισσότερο. Έχουμε δημιουργήσει μια διευθυντική ομάδα στο EMI που ασχολείται μόνο με τον καρκίνο, είναι καινούριο αυτό. Τώρα οι επιχειρήσεις βλέπουν ότι είναι μεγάλο πλεονέκτημα το να συνεργάζονται για τέτοιου είδους ασθένειες. Επίσης η ρομποτική μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα, ένα από τα σχέδια στα οποία αναφέρθηκα έχει οδηγήσει στη δημιουργία στην Ολλανδία μιας ρομποτικής δομής υψηλού επίπεδου με υψηλό κόστος εκπαίδευσης και κατασκευής, αλλά αυτό έχει δημιουργήσει επίσης και πολλές θέσεις εργασίας υψηλού επίπεδου. Ε, δεν ασχολούμεθα πάρα πολύ με τα θέματα της ορθοπαιδικής και των ε, πρόσθετων μελών, αλλά ε, με θέματα προχωρημένων μορφών θεραπείας. Είναι κάτι το οποίο καλύπτει κυρίως τις σπάνιες ασθένειες, σπάνιους καρκίνους, αλλά είναι κάτι που στο μέλλον μπορεί να διευρυνθεί και σε άλλες ασθένειες. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει ο πρόεδρος Μπούζεκ. Τα θέματα αυτά πράγματι επηρεάζουν την κοινή γνώμη και θα θέλαμε να γνωρίζουμε γιατί το IMI και άλλες τέτοιες προσπάθειες μπορεί να παίξουν σημαντικό ρόλο και να χρησιμοποιήσουν σωστά τα χρήματά μας για τον ορίζοντα 2020. Εμείς ασχολούμεθα κυρίως με την αρχή της προσθετικότητας. Προσπαθούμε να δούμε τι είναι αυτό το οποίο δεν θα γινόταν χωρίς το IMI. Η οργάνωσή σας λειτουργεί με έναν απλά τυπικό συνεργατικό σε εισαγωγικά τρόπο. Εμάς μας ενδιαφέρει για το πώς θα μπορέσουμε να εξηγήσουμε στους ε, ε, πολίτες τους εκλογής μας το ενδιαφέρον του εγχειρήματός σας. Κοιτάξτε, τρία πράγματα, τρία επιχειρήματα. Πρώτον, είναι μια πρωτοβουλία όπου για πρώτη φορά οι εταίροι βιομηχανικοί συνεργάζονται μεταξύ τους. Μιλάμε για τη φαρμακευτική βιομηχανία, η οποία είναι ιδιαίτερως ανταγωνιστική. Τώρα βλέπουμε για πρώτη φορά 7, 8, 9 επιχειρήσεις να συνεργάζονται. Ε, στην ουσία ορίζουν κάποιες προκλήσεις και κάποιες δυσκολίες τις οποίες θεωρούν ότι μόνες τους δεν θα το καταφέρουν να κάνουν. Χρειάζονται την δημιουργικότητα και των μικρομεσαίων και των πανεπιστημιακών ακαδημαϊκών ερευνητικών κέντρων. Και εμείς μπορούμε να λειτουργήσουμε σε επίπεδο κλίμακας λόγω του συνδυασμού των πόρων και από πλευράς της ε, ε, του ιδιωτικού τομέα και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κάποιοι συνάδελφοι στις Ηνωμένε Πολιτείε και την Ασία ε, ζηλεύουν θα έλεγα την κλίμακα στην οποία μπορούμε να εργαστούμε πλέον. Ε, σας εύχομαι να συνεχίσετε μια εικονοποιητική λοιπόν προσπάθεια και ελπίζουμε στο μέλλον να υπάρξουν και αντίστοιχες ε, συνδυαστικές προσπάθειες, κοινέ προσπάθειες σαν τη δική σας. Κοιτάξτε συνάδελφοι, πάμε στο τελευταίο σημείο για σήμερα το πρωί είναι το σημείο 6 ε, ενημέρωση από τους συνεχιζόμενους τριμερείς ε, διαλόγους έχουμε έναν πολύ σημαντικό ε, ενεργειακή αποδοτικότητα και σήμανση πάνω σε θέματα τέτοιας ενεργειακής αποδοτικότητας. Ίσως να μην είναι τόσο εύκολο το θέμα αυτό, αν και είναι σημαντικό και γι' αυτό θα ακούσουμε με προσοχή τον κύριο Ντάριο Ταμπουράνο. Έχετε το λόγο κύριε Ταμπουράνο. Ο τριμερής διάλογος αφορά πρόταση κανονισμού για την αναθεώρηση των κριτηρίων της ετικετοθεσίας όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση για διάφορα προϊόντα μεταξύ των οποίων είναι και τα πιο αγνωστά πλυντήρια, ψυγεία και όχι μόνο ε, αφορά θερμάστες, ε, περιβαλλοντικούς ε, συσκευές θέρμασης κλπ. Όπως γνωρίζετε, θα θυμόσαστε στην Ολομέλεια, ψηφίστηκε η θέση του Κοινοβουλίου με πολύ ικανοποιητική πλειοψηφία θα έλεγα. Στους ακόλουθους τριημερείς διαλόγους ελπίζαμε να ολοκληρώσουμε την προσπάθεια σε τρεις συναντήσεις. Δυστυχώς δεν έγιναν τα πράγματα. Υπάρχουν προβλήματα που σχετίζονται με τα διάφορα άθρα θεσμικής φύσεως που ξεπερνούν το χαρτοφυλάκι αυτό, το θέμα των εξουσιοδότησης πράξεων και των εκτελεστικών πράξεων. Πέρσι, ε, στο το Συμβούλιο κατέληξε σε θέση όσον αφορά το θέμα αυτό ε, θέτοντα τα πάντα στι κατεξουσιοδότηση πράξη και τι εφαρμοστικέ πράξει. Η θέση του Κοινοβουλίου προβλέπει τι κατεξουσιοδότηση πράξη. Υπήρξε διοργανική συμφωνία ε, πάντα το περσινό χειμώνα που ερμηνεύεται όπως από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή Συμβουλίου και Κοινοβουλίου όσον αφορά τις διαδικασίες που πρέπει κανονικά να ακολουθούνται όσον αφορά το Better Legislation το Συμβούλιο παραμένει σταθερό στη θέση των εφαρμοστικών πράξεων και το Κοινοβούλιο παραμένει σταθερό στη θέση των κατεξουδότησης πράξεων. Εάν δεχόμαστε τις εφαρμοστικές ε, ε, πράξεις θα μπορούσε να μπλοκάρει το όλο θέμα στη διάσκεψη των Πρόεδρων. Αυτό πέρα το περιεχόμενο του χαρτοφυλακίου είναι ένα θέμα που μπορεί να παρουσιαστεί σε κάθε νομοθετική πράξη που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Τώρα όσον αφορά το περιεχόμενο, ε, είναι πολύ τεχνικής φύσεως το θέμα, δεν θα μπω σε βάθος των άρθρων. Ε, ουσιαστικά διαφαίνεται η δυνατότητα συμφωνία στα κρίσιμα θέματα ή κλι, η η, το, το, η μέγεθος των νέων ετικετών, το rescaling, θέμα χρονοδιαγράμματος για το rescaling και η έννοια του rescaling, Όσον αφορά την database, τη βάση δεδομένων, ε, είμαστε πολύ κοντά. Σε συμφωνία υπάρχουν και άλλα θέματα ίσονο σημασία. Η ενίσχυση τη ε, αγορά για την αγορά και η προστασία του καταναλωτού σε περίπτωση ε, προβληματικού προϊόντο και αποζημιώσεω, που αυτά μπορούν να αντιμετωπιστούν. Το πρώτο νομοθετικό χαρτοφυλάκιο που είναι σημαντικό μετά το σκάνδαλο τη Volkswagen που έδειξε τα κενά κάποιων κανόνων που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε στη διάθεση ε, των συναδέλφων για ειδίποτε ερώτηση να απαντήσω. Ευχαριστώ τους συναδέρφους και βέβαια ευχαριστώ τον Πρόεδρο που πάντα ήταν στο πλευρό μας και στη συνεδρίαση των σκιωδών και κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο. Σας ευχαριστώ εκ νέου. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σιγητά, ευχαριστώ Ντάριο Ταμποράνο. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα, δεν είναι εύκολες οι διαπραγματεύσεις που έχουμε μπροστά μας. Στον επόμενο γύρο δεν ολοκληρώσαμε σε τρεις γύρους συνομιλιών, αυτό το είπε και ο κ. Σταμπουράνο. Υπάρχουν ερωτήσεις, σχόλια ενδεχομένω ως σχετικά με αυτά που είπε ο εισηγητής μας. Από τη δική μου πλευρά, αν επιτρέπετε, θέλω να πω μόνο ένα πράγμα. Είναι σημαντικότατο να πετύχουμε, πώς να το πω, κάτι σαν μια κοινή θέση ούτως υπήν του Ευρωκοινοβουλίου. Γιατί το λέω αυτό. Διότι βέβαια η εντολή που ψηφίσαμε στην Ολομέλεια πρέπει να αλλάξει κάπως. Όπως γνωρίζετε στις διαπραγματεύσεις δεν μπορούμε να πετύχουμε αυτά που θέλαμε και προτείναμε στην Ολομέλεια ή στην Επιτροπή μας. Αυτό είναι προφανέστατο. Άρα θα ήταν πολύ καλό εάν ακόμα και πριν τη συνεδρίαση τεχνικού επίπεδου την Παρασκευή οι σκιώδεις εισηγητές μας και ο εισηγητής αν μπορούσαν να συναντηθούν να δουν τι είναι εφικτό από τη δική μας πλευρά. Το Συμβούλιο προτείνει κάποιες λύσεις και θα πρέπει να είναι αρκετά ξαφές αν είμαστε έτοιμοι να συμφωνήσουμε. Βέβαια πρέπει να υπερασπιστούμε τη θέση μας. Αυτό είναι προφανές. Όλοι το γνωρίζουν. οι σκιώδεις εισηγητές και ο εισηγητής μας αυτό προσπαθούν να κάνουν. Από αυτή την πλευρά δεν έχουμε πρόβλημα. Μια ισχυρή κοινή θέση επί του θέματος κάτι εντελώς διαφορετικό, ε, κάτι που υπερασπιζόμαστε από κοινού και εγώ το με υπερασπίζω αυτή τη θέση, είναι κάτι εντελώς διαφορετικό το εξή, ότι η κατεξουσιοδότηση πράξη είναι απαραίτητη στη συγκεκριμένη περίπτωση, όχι εφαρμοστική πράξη. Το ίδιο ισχύει και στον πρώτερο κανονισμό. Και ήταν αναμενόμενο μετά την τελευταία μας συμφωνία με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για καλύτερη διαδικασία νομοθεσίας. Ας ακολουθήσουμε λοιπόν αυτή την κατεύθυνση. Κατεξουσιοδότηση πράξη και όχι εφαρμοστική. Όπως είναι η θέση του Συμβουλίου, επιθυμία του Συμβουλίου και πρόταση του Συμβουλίου. Εάν δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, και τα πάντα είναι λίγο πολύ σαφή για σας. Εγώ θα έλεγα ότι μπορούμε να ολοκληρώσουμε την πρωινή μας συνεδρίαση. Όχι το πρωί βέβαια, αλλά το απόγευμα. Καλά είμαστε. Θα ολοκληρωθεί το απόγευμα. Τα πάντα είναι ωραία και καλά. Ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε στις 3. Πολύ σημαντική πληροφορία. Στις 9 το πρωί, αύριο, ψηφοφορία. Τρίωρη ψηφοφορία. Αυτό προβλέπει η γραμματεία. Μαζί με το διάλειμμα που θα χρειαστεί, ας πούμε 3,5 ώρες. Είστε έτοιμοι λοιπόν για πολύ σκληρή δουλειά. Στην Επιτροπή είτε εργαζόμαστε πάρα πολύ σκληρά. Υπέροχη, φοβερή επιτροπή. Στις 3 λοιπόν σήμερα και αύριο το απόγευμα έχουμε κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή Πολιτισμού. Πολύ σημαντικό και αυτό. Δημιουργική βιομηχανία. Μια νέα ιδέα, αρκετά νέα, που αναπτύχθηκε στη δική μας ε, Επιτροπή. Σας καλώ λοιπόν και ολοκληρώνουμε τις εργασίες αύριο στις 6.30, όχι σήμερα, 6.30 αύριο. Όλοι θα είναι παρόντες, εγώ θα είμαι παρόν. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, θα τα πούμε στις 3, καλή όρεξη.